Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ε, αν θέλετε να καθίσετε. Θα χρειαστείτε βέβαια και τις ε, κάρτες σας για ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάμε λοιπόν με το σημείο υπαριθμών 10 της ημερήσια διαταξής ε, για, τις, ε, για τους ισχυρισμού υγείας ε, και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στην κυρία Γανάτε Ζώμα η οποία θέλει να κάνει μια δήλωση εκ μέρους του ΕΛΚ η οποία επιθυμεί και να γραφτεί στα πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια δήλωση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ε, το θέμα αυτό και σχετικά με το βέτο για τον κατάλογο των ισχυρισμών υγείας. Το συζητήσαμε επανειλημμένα και τελικά αποφασίσαμε να δώσουμε ένα μήνυμα στην Κομισιόν και να συμφωνήσουμε με το ΒΕΤΟ. Θα ήθελα λοιπόν να καταθέσω μια γραπτή δήλωση στα πρακτικά. Την έχω προετοιμάσει, μπορώ να τη δώσω ε, στη γραμματεία αν θέλετε μπορείς να τη, μπορώ και να τη, στείλω ηλεκτρονικά. Ε, ο κατάλογος αυτός ε, μας δημιουργεί πολλές επιφυλάξεις και αυτές τις επιφυλάξεις τις εκφράσαμε χθε στη συζήτηση. <clears throat> Θα ήθελα λοιπόν να δηλώσω ότι εμείς δεν επιθυμούμε να στραφούμε κατά της ΕΦΣΑ και των αποφάσεών της. Τον αντίον είμαστε υπέρ της ΕΦΣΑ και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης της, αλλά τελικά φαίνεται ότι η ΕΦΣΑ δεν είναι αρμόδια για διαφημιστικά σποτ. Ε, Εμείς θέλουμε η Κομισιόν να μας λάβει σοβαρά υπόψη της. Ε, γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό που σας είπα και δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αγνοεί το Κοινοβούλιο με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις αγνώντας μας πλήρως και κυρίως ε, τη στιγμή που επίκειται μια διαδικασία σκρούτινη. Πρόκειται για τα διατροφικά προφίλ τα οποία ακόμα δεν έχουν οριστεί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μόνη τις πολιτικές αποφάσεις επίσης ε, να ε, προκαταλάβει τα διατροφικά προφίλ και ως εκ τούτου <clears throat> ανακατανέμει και ανασυντάσει τον κατάλογο ε, και γι' αυτό το λόγο εμείς δεν συμφωνούμε και κατόπιν τούτου θα ψηφίσουμε αρνητικά παρότι βέβαια όπως σας είπα θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά της παραπλανητικής διαφήμισης και αυτό νομίζω αποδεικνύεται και από τον τρόπο που λειτουργήσαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτή λοιπόν τη δήλωση θα την καταθέσω στα πρακτικά. Επιθυμεί παρακαλώ κάποιος να διαφωνήσει από ό,τι βλέπω δεν ισχύει ως εκ τούτου μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, με, τον, ε, με την ψηφοφορία. ψηφίζουμε για το παράρτημα σχετικά με τα τρόφιμα. Και προτείνω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία έκλεισε η ψηφοφορία. 22 υπέρ, 37 κατά και μία αποχή. Ευχαριστούμε πολύ. Απορρίπτεται. Ε, πάμε τώρα. Πάμε στην έκθεση Γκεμπραντή. Στρατηγική διοπικιλότητας ε, για το 2020. Hier haben Bring eine Πρόκειται για ένα χοντρό πακέτο, όμως ε, έχουμε και πολλές ε, συμπυκνωμένες τροπολογίες. Consolidated Amendment 1. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 2, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Πάμε στην 3, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τέσσερα, παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την επόμενη, την 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 6 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθυμών 7. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 9. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για τη 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για την 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 13. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για τη συμβαστική υπαριθμών 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπερτιμών 26. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία υπερτιμών 36. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 και 39 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την ε, τροπολογία 38 σε τμήματα. Ποιος να παρακαλώ υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία ε, της Επιτροπής Περιφερειών. ένα, Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 42 σε τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αλλά ηλεκτρονική επαλήθευση για την 42, για το πρώτο τμήμα, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία, 36 υπέρ, 26 κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, Πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 33 υπέρ, 29 κατά. Κατοπιν τούτου εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την ΙΤΡΕ 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αγκρι 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για την 49. Πάμε κατόπιν, κατόπιν τούτου στη 48. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την τροπολογία 50 σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Κατά, με τώρα κατά. Αποχές ε, μπορούμε να ξαναψηφίσουμε για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 38 υπέρ, 23 κατά αν σηκώνετε όλοι σωστά το χέρι σας, νομίζω τα πράγματα θα είναι πιο απλά. Απευθύνομαι στους συντονιστές κυρίως. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 53. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για την 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για την 9 της Επιτροπής Αλίας υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση για την 9 της Αλίας. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. τους φιλελεύθερους υπάρχει ένας που είναι επιπλέον είναι περισσότεροι κατά ένα οι φιλελεύθεροι. Ε, πρόεδρε, δεν νομίζω ότι μπορείτε να το σχεριστείτε πολύ συχνά αυτό για μένα. Η ιδέα του να, είναι, να περισσεύουν οι φιλελεύθεροι, αυτό ομολογώ ότι μάλλον σπανίζει. Κλείνει λοιπόν η ψηφοφορία. Παρακαλώ να σηκώνετε σωστά το χέρι σας, γιατί δεν θα υπάρχει πλέον ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε για την Ήτρε Νέα. Υπέρ παρακαλώ. Ποιο είναι υπέρ τη Ήτρε Νέα. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. Ήτρε 10. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα της Ήτρε 10. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές και αυτή εγκρίνεται. Πάμε στην Ήτρε 11. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ρέγγι 4 ε, όμως ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την ήτρε 22 ψηφίζουμε παρακαλώ ψηφίσατε όλοι Έκλεισε η ψηφοφορία. 30 υπέρ, 33 κατά, απορρίπτεται. Πάμε στη Ρέγγι 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 20, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, Ξαναψηφίζουμε. Ήτρε 20, πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 20 για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 2. Υπέρ κατά, αποχές ε, γκρίνεται Τροπολογία 63, υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. 64, υπέρ, κατά, αποχές, ε, παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε για την 64. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Ένας παραπάνω στο ΕΛΚ. Λοιπόν, 33 υπέρ, 30 κατά, εγκρίνεται. Τώρα, ψηφίζουμε για την 65. Υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, ε, ε ψηφίζουμε για την 65. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 32 υπέρ, 31 κατά. Κατόπιν τούτου εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την 66. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 67 σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την Ήτρε 3, πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, ε, αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για το δεύτερο τμήμα της ΙΤΡΕ 3. Έκλεισε η ψηφορία. 34 υπέρ, 28 κατά, κατοπιν τούτου εγκρίνεται. Ρέγγι 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 68 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ε, παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε για την 68 ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι έκλεισε η ψηφοφορία 30 υπέρ 33 κατά κατόπιν τούτου απορρίπτεται τώρα Ψηφίζουμε για την 69. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 69. ...32 υπέρ, 31 ε, κατά, ε, μόλις που εγκρίθηκε, οριακά. Τροπολογία 70. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 77. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές Ποιος είναι υπέρ της 77 κατά αποχές. Νομίζω είναι σαφές το αποτέλεσμα. Τώρα ψηφίζουμε για την 79. Έκανε λάθος ο πρόεδρος. 79. Εστέρντε Λάγκε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 6. Υπέρ. Κατά Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την ΙΤΡΑ 6. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Η 80 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για την 81 σε τρία τμήματα. Για το πρώτο τμήμα παρακαλώ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για το δεύτερο τμήμα υπέρ, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Για το πρώτο τμήμα της 81. Έκλεισε η ψηφορία. 31 ε, υπέρ, 32 ε, κατά. Πάμε στο δεύτερο τμήμα για το δεύτερο τμήμα, ποιο είναι παρακαλώ υπέρ της ε, τροπολογία 81, υπέρ κατά, αποχές, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε για την 81 και το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφορία. 42 ε, υπέρ, 21 κατά, Μπερδεύουμε λιγάκι με το ότι έχετε αλλάξει θέση στην αίθουσα. Τέλος πάντων, ψηφίζουμε τώρα για το τρίτο τμήμα, για το τρίτο τμήμα της 81, παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για την 82, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέγγι 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την 85 σε τρία τμήματα. Παρακαλώ ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Για το τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση για το τρίτο τμήμα της 85. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 32 <clears throat> υπέρ, 30 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την 116. Υπέρ παρακαλώ. ...116 καταπίπτει... ...οπότε ψηφίσουμε την Άγκρη 18 υπέρ... ...κατά... ...αποχές εγκρίνεται... Ρέγγι 13. Ε, υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 2. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 86 υπέρ 86 υπέρ αποχές απορρίπτεται οπότε περνάμε στην 103 ποιος είναι υπέρ της 103 παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται 46 τροπολογία υπέρ κατά Αποχές. Ψηφίζουμε την 46. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. 24 υπέρ, 35 κατά, οπότε απορρίπτεται. Ρέγγι 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105. Α, θα ελέγξουμε την 106. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Ισοψηφία 31. Απορρίπτεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, καταπίπτει. Εφόσον εγκρίθηκε 105. Σαφές. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά. αποχές να κάνουμε έλεγχο. Ψηφίζουμε την 109. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 32 υπέρ, 29 κατά, εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ή 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 7 υπέρ αποχές, ε, κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 112 καταπίπτει. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές ασαφές να ελέγξουμε 118 ηλεκτρονικά Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 46 υπέρ, 14 κατά. Δεν, ήταν, δεν φαινόταν καθαρά από εδώ στο Προεδρείο. Παρά τη μεγάλη διαφορά. 120, 121 συγγνώμη, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε τώρα στην 138 όπου έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 5 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε αρκετές αρκετές Και περνάμε στην τροπολογία 155. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και πάλι περνάμε αρκετές. Άγκρι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα 180 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 181 υπέρ κατά άλλη μια φορά παρακαλώ 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 α θα ελέγξουμε την 181 181 ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίσατε όλοι πέρας 35 υπέρ 25 κατά εγκρίνεται Λοιπόν, μα μόλις ελέγξαμε την 181 και ηλεκτρονικός. Α, μάλιστα. Ορισμένοι κατάλαβαν 182. Οπότε ξαναρχίζουμε. Ξαναψηφίζουμε την 181 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 37 υπέρ. 24 κατά. Ωραία. Πολύ ωραία. 182. 182. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Α, αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 184 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 185 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 186 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Περνάμε και πάλι αρκετές και περνάμε στην 197 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ. 198. 198 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 199 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. 199. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 200 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές ασαφές άλλη μια φορά 201 υπέρ παρακαλώ το χέρι ψηλά υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ασαφές. 201. Ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. 18 υπέρ, 44 κατά. Αλλά δεν φαινόταν από εδώ. Παρακαλώ, ε, αν σηκώνετε καλά το χέρι, μας διευκολύνεται. Άγκρι 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 16 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 204 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος 202 παρακαλώ ψηφίσατε όλοι πέρας ισοψηφία με, με 30 απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...208... ...δύο τμήματα... ...πρώτο... ...υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...εγκρίνεται... ...δεύτερο τμήμα... ...υπέρ... ...κατά... ...αποχές... Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 212 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πες 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πες 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 216 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Λοιπόν, παρακαλώ έλεγχο στο πρώτο τμήμα της 2.16. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 40 υπέρ, 22 κατά. Σας παρακαλώ να σηκώνετε καλά το χέρι, δεν είναι σαφές. Δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα της 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 218 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.20 καταπίπτει. 2.22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.23 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 5 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί ούτε η 8, ΠΕΣ 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΠΕΣ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΠΕΣ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΠΕΣ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάλι περνάμε αρκετέ και περνάμε στη 2.33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 3, ρέγγι, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.46, κατά τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Α, καταπίπτει. 2.47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.53 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτε, δεύτερο τμήμα της 253 υπέρ. Α, καταπίπτει. Περνάμε λοιπόν στο τρίτο τμήμα της 253 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται 2.55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ρέγγι 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 259 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 260 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 261 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 262 υπέρ. Κατά άποχες. Δεν είναι σαφές. Να ελέγξουμε. 262. 262 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 31 υπέρ, 30 κατά. Εγκρίνεται. 263 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχέ, Εγκρίνεται. Ήτρε 17 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ήτρε 18 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Υπέρ του τρίτου. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 264 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέγγι 10 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί 267 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πέσω 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 268 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 269 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές ασαφές ηλεκτρονικός έλεγχος. 269. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 31 υπέρ 29 κατά εγκρίνεται. 2,70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2,71 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 2,72 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 2,73 υπέρ. Κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος. 2.73. Άρχεται για τη 2.73. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 32 υπέρ. 29 κατά εγκρίνεται. Να περάσουμε τώρα στη 2.82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2.83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 2.85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.86 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές και το ε, δεύτερο εγκρίνεται ρέγγι 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ρέγγι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ρέγγι 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, σκέψει σκέψεις τώρα λοιπόν τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έχουμε δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, τη 2 και 3, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές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 αποχές για να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 29 υπέρ. 33 κατά. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και να κάνουμε την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά Άρχεται η ηλεκτρονική συνολική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ακόμη δύο δεν έχουν ψηφίσει. Ψηφίσατε όλοι. 58 υπέρ. Κανείς κατά. Τέσσερις αποχές. Θερμά χαρακτήρια για τον Γιάνν Γκέρμπερ και Μπράντι για αυτή την έκθεση. Θαυμάσια.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 που παρασκευάζει η γαλλική εταιρεία PIP. Ποιο θέλει να ψηφίσουμε, να σηκώσει παρακαλώ το χέρι. Κατά, αποχές. Έτσι λοιπόν αυτή η προφορική ερώτηση εγκρίθηκε ομόφωνα και πάμε τώρα στη συζήτηση. Der Kollege Ο συνάδελφο Όλμαν. Ε, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι. Εδώ λοιπόν πρόκειται για το εξής. Υπάρχει αυτό το σκάνδαλο για τα εμφυτεύματα στήθου τη εταιρεία PIP. Εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα και πιο συγκεκριμένα καλούμε την Επιτροπή τις προτάσεις μας ε, που τις ε, αναφέρουμε σε 7 σελίδες. Ε, τις προτάσεις μας αυτές να τις συμπεριλάβει στην αναθεώρησή της, στην αναθεώρηση σχετικής οδηγίας. Και είναι σαφές ότι η οδηγία αυτή λειτουργεί ικανοποιητικά. Αποδείχθηκε ότι η εταιρεία αυτή αναπτύσσει εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι τώρα μπόρεσε να ε, ξεφύγει. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε αυστηρότερους ελέγχους, ε, χρειαζόμαστε ε, τη δυνατότητα να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα εκ των υστέρων τις πρακτικές, αλλά χρειαζόμαστε και τις τεχνικές εκείνες οι οποίες θα μας επιτρέπουν να ελέγχουμε τα προϊόντα με μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι το πράξαμε μέχρι σήμερα. Και από όλη αυτή την πρακτική συνάγουμε επίσης ότι το μέχρι τώρα σύστημα έχει μία χίλιο πτέρνα με την εξής έννοια ότι εξετάζει θέματα κατασκευής. Αυτό λοιπόν έγινε γραπτά χωρίς να εξεταστεί το συγκεκριμένο προϊόν. Ε, πρέπει να το δούμε λιγάκι. Θα πρέπει να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι σε συγκεκριμένα προϊόντα. Σε εθνικό επίπεδο βεβαίως ε, είναι σκόπιμο να έχουμε ένα μητρό εμφυτευμάτων έτσι ώστε σε περίπτωση αμφιβολίας να μπορούμε να δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Δεν πρόκειται τώρα μόνο για αυτή την εταιρεία, την ΠΕΙΠΕ, αλλά ε, μιλάμε και για άλλα εμφυτεύματα, εμφυτεύματα ισχύου, τα οποία και αυτά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα ε, λόγω του μετάλλου που περιλαμβάνεται στα εμφυτεύματα αυτά. Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και νομίζω επίσης ε, ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την προστασία των δεδομένων λέγοντας ότι αν ένας ε, άμεσα αν ένας ασθενής διαφωνεί ριζικά, δεν πρέπει απαραίτητα να ανακοινώνεται το όνομά του. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η Κομισιόν θα προετοιμάσει ε, την οδηγία, τη σχετική οδηγία, λαμβάνω τις υπόψη αυτά που είπα και χαίρομαι για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Η Λίντα Μακάφνη έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε τον Ιανουάριο μία πάρα πολύ μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, μίλησε ειδικότερα για την οδηγία για τα ιατροτεχνικά ε, βοηθήματα, Τώρα γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νέα νομοθεσία, κάτι το οποίο δεν ήταν σαφέ στην προηγούμενη συζήτηση. Ούτω ή άλλω θα το ψηφίσουμε αυτό στην ε, Ολομέλεια το Μάιο. Επαναλαμβάνουμε αυτά που είπαμε τον Ιανουάριο δηλαδή, ότι χρειαζόμαστε την αναθεώρηση της ε, νομοθεσίας. Θέλουμε ένα μητρό για τα εμφυτεύματα στήθους και τα άλλα εμφυτεύματα σε κάθε χώρα. Ε, έχουμε, όχι, μόνο έχουμε χιλιάδες ε, γυναίκες με εμφυτεύματα στήθους που ανησυχούν, αλλά έχουμε και χιλιάδες γυναίκες που δεν ξέρουν και τι είδους εμφυτεύματα έχουν. Και αν είχαμε λύσει το πρόβλημα αυτό με το Συμβούλιο πριν από 10 χρόνια, δεν θα είχαμε το ίδιο πρόβλημα, δεν θα το πρόβλημα αυτό σήμερα. Εντάξει, υπάρχει η γραφειοκρατία, αλλά υπάρχει και το θέμα τη προστασία των πολιτών που είναι πολύ σημαντικότερο. Πρέπει λοιπόν το Μητρό να αποτελέσει τμήμα τη νομοθεσία. Ελπίζω λοιπόν ότι το Συμβούλιο θα μα υποστηρίξει. Θα μα υποστηρίξει, εκπροσωπείται σήμερα εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία. Γιατί από τότε που έγινε η συζήτηση για το θέμα αυτό υπάρχει ένα νέο θέμα με τα εμφυτεύματα ε, ισχύων ε, και σε μερικές χώρες και αναρωτιέμαι ε, αν υπάρχουν νεότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα των εμφυτευμάτων ισχύων γιατί υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία που έχουν αλλάξει ε, σε σχέση με τα εμφυτεύματα των ισχύων και ίσως θα έπρεπε να έχουμε καλύτερες ε, κλινικές δοκιμές των εμφυτευμάτων πριν ε, τοποθετηθούν στην αγορά ευρέως. Γιατί κάποιοι Βρετανοί πολίτες θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα εμφυτεύματα αυτά λόγω του σχεδιασμού τους. Οπότε θα ήθελα να ακούσω τι θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε τις νομοθετικές αλλαγές που χρειαζόμαστε. Äh, Ο συνάδελφος Τζιλ Πανιό, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για ένα ψήφισμα το οποίο Εκτός από τις δυσκολίες ε, που ε, συναντήσαμε ε, με τα εμφυτεύματα στήθους εταιρεία PayPay, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο λοιπόν ε, διαπιστώνουμε μέσω του ψηφίσματος αυτού ότι η μεταγραφή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ε, για τα ιατροτεχνικά σκευάσματα και βοηθήματα δεν ε, παρεμπόδισε αυτήν την υγειονομική απάτη. Αυτό είναι το πρώτο που διαπιστώνουμε στο ψήφισμα αυτό. Το γεγονός αυτό μάλιστα έδειξε μια δυσλειτουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μέλων και της διεθνούς όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, όπω επίση και έλλειψη χνηλασιμότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα ιατροτεχνικά βοηθήματα. Το ψήφισμα διαπιστώνει επίση την αποτυχία του τρέχοντο συστήματος ε, πιστοποίησης και ελέγχων και ε, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα του να ληφθεί υπόψη αυτή η απάτη στην αναθεώρηση της οδηγίας για τα ιατροτεχνικά βοηθήματα, όπως μόλις είπε η ε, προλαλήσα σας συνάδελφος η κυρία Μακάβαν. Βλέπουμε ότι υπό το φως όσων συνέβησαν ε, με τα εμφυτεύματα της εταιρείας ΠΕΙΠΕ και άλλα ιατροτεχνικά βοηθήματα, σήμερα είναι στην επικαιρότητα τα οποία μάλιστα δημιουργούν σοβαρές δυσλειτουργίες ε, στην υγεία και μιλάω για τα εμφυτεύματα ισχύων ε, που ήταν ε, που δημιούργησαν μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά το περιεχόμενο, τα συστατικά τους. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το εν λόγω ψήφισμα και για να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της νέας ε, ε, πρότασης ε, που έχει δρομολογηθεί για τα ιατροτεχνικά βοηθήματα να μας υποβάλει προτάσεις οι οποίες θα είναι υποχρεωτικές για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους καταστάσεις στο μέλλον. Θα ήθελα επίσης να κάνω και μία πρόταση, θα υποβάλω και σχετική τροπολογία, ώστε οι κατασκευαστέ ιατροτεχνικών βοηθημάτων όπως τα εμφυτεύματα στήθους για παράδειγμα, να είναι υποχρεωμένοι, κάτι που δεν ισχύει σήμερα, να αναφέρουν αν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος εγκατάστασής τους, υπάρχει μία διαδικασία ε, που να έχει ξεκινήσει ε, γιατί ε, δεν μας υποχρεώνει, δεν μας ε, εμποδίζει κανείς να δεν υποχρεώνει κανείς να ενημερώνει ο κατασκευαστής ε, τις ε, αρχές της χώρας μέλους στην οποία βρίσκεται, αλλά δεν εμποδίζει και να ενημερώσει τους, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, όπως έγινε για παράδειγμα με την γαλλική εταιρεία Paper, ε, γιατί υπήρξαν περιπτώσεις και σε άλλα κράτη-μέλη. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι φιλελεύθεροι ε, επικροτούν το ψήφισμα. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ εξισορροπημένο και καλύπτει ε, πολλά ζητήματα ε, που πρέπει να εξεταστούν ε, κατόπιν της συζήτησή μας τον Ιανουάριο και της κατάστασης με την ΠΕΙΠΕ. Υπάρχει μια διαδικασία απάτης, την οποία, ε, η οποία διερευνάται στην Καλία. Υπάρχουν πολλά παραθυράκια στους νόμους και πιστεύουμε ότι πρέπει πραγματικά να γίνει αναθεώρηση του πλαισίου για τα ιατροτεχνικά βοηθήματα αυτό είναι ε, το μάθημα που πρέπει να πάρουμε και πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι όλα τα βοηθήματα ίδια τα ιατρικά και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση κινδύνου ε, κατά περίπτωση. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, όλοι ο Πρόεδρος. Κυρία Κούκουβιτς. Ευχαριστώ, κύριε Κύριε Πρόεδρε, εγώ χαιρετίζω αυτό το ψήφισμα. Παράλληλα όμως λυπάμαι πάρα πολύ που φτάσαμε μέχρι εκεί. Λυπάμαι πολύ που συνέβη αυτό σε τόσες πολλές γυναίκες οι οποίες ε, κατέστησαν θύματα της ε, ε, βεβαιασμένων επεμβάσεων και παραλήψεων. Πρέπει να τονίσουμε το θέμα της αριστείας της, των βέλτιστων πρακτικών, γιατί υπάρχουν προϊόντα ε, τα οποία για να έρθουν σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα πρέπει να καλύπτουν υψηλότατες προδιαγραφές. Άρα δηλαδή οφείλουμε να απευθύνουμε έκκληση στην ε, ιατρική η οποία παράγει αυτά τα προϊόντα. Η αριστεία λοιπόν, αυτό είναι το καθοριστικό θέμα. Το πρόγραμμα Horizon τονίζει κάτι τέτοιο. Ε, βεβαίως ε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ενημερώνονται οι νέοι. Απευθύνομαι κυρίως στους νέους γιατί πολλοί εξ αυτών έχουν έμονες ιδέες, ιδεολειψίες, νέες γυναίκες, οι οποίες ε, διατρέχουν όλους αυτούς τους κινδύνους με τέτοιου είδους εμφυτεύματα. Οφείλουμε λοιπόν να απευθυνθούμε και στη βιομηχανία αλλά και στην κοινή γνώμη. Να ενημερώσουμε καλύτερα για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα εμφυτεύματα κυρία Κουντάκη, εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Και εγώ ε, χαιρετίζω... Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ε, χαιρετίζω το ψήφισμα. Ελπίζω με την αναθεώρηση της οδηγίας να καλύψουμε αρκετά, αρκετούς τομείς. Ε, μιλούμε για απάτη στην περίπτωση της εταιρείας PayPal, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε ευρύτερα ζητήματα σε σχέση με τα εμφυτεύματα και άλλα κομμάτια που ε, τοποθετούνται στο σώμα ε, δεν με έχουν ε, πείσει ορισμένα πράγματα. Καταλαβαίνω την ανάγκη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει το μητρό. Προφανώς το νοσοκομείο πρέπει να ξέρει ποιον έχει εγχειρήσει, Τώρα, πώς είναι δυνατόν να τηρήσουμε ένα εθνικό μητρό και να το ενημερώνουμε. Ο κόσμος μετακινείται, αλλάζει διευθύνσει, ο κόσμος ε, φεύγει από τον κόσμο αυτό, οπότε πώς είναι δυνατόν να ε, τηρήσουμε αυτό το μητρό. Με, απασχολεί, λοιπόν, με απασχολούν οι λεπτομέρειες. Μου αρέσει όμως το θέμα του διαβατηρίου γιατί ακριβώς αυτό δίνει, ιδιαίτερη, δίνει βαρύτητα στον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να μετακινείται και το παίρνει μαζί του. Ενώ αντίθετα το μητρό ε, σε συνδέει με την εθνική σου ασφάλεια και ε, δημιουργείται μια κοινωνία του ε, μεγάλου αδερφού κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι τα ζητήματα της οδηγίας για τα ιατροτεχνικά βοηθήματα πρέπει να καλυφθούν και ελπίζουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία λοιπόν. Ε, έκλεισε ο κατάλογος των ομιλητών. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ζακλίν Μινό, ε, η οποία είναι διευθύντρια από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, γιατί ετέθησαν ερωτήματα που ενδεχομένως καλά θα ήταν απαντήτων. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, εκτενέστατη απάντησή σας σε αυτές τις γραπτές ερωτήσεις που είχαμε υποβάλει. Υπάρχουν όμως ε, και άλλες ερωτήσεις. Ε, συνάδελφος Σίλντας και η κυρία Λένα Μακέβν. Παρακαλώ, Σίλντας. Ή συνάδελφος Σίλντας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τους άλλους ομιλητές ε, για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έλαβα χώρα. Ε, κοιτάξτε, στη δική μου τη χώρα υπήρξαν πολλές περιπτώσεις ε, αιτήματος αποζημίωσης ατόμων που αντιμετώπισαν προβλήματα με τα εμφυτεύματα τα, της εταιρεία PEP. Αυτό συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, τα εμφυτεύματα ισχύου και ρωτώ λοιπόν, μήπως είναι δυνατόν στο πλαίσιο της οδηγίας ε, να προταθεί να υπάρξει ένα ταμείο ε, το οποίο θα αποζημιώνει ε, τους ανθρώπους όταν υποστούν ζημιά είτε όταν έχει πάυσει τη δραστηριότητά του ο κατασκευαστής είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν σε συνδυασμό με την ταξινόμηση αυτών των προϊόντων στην αγορά. Γιατί νομίζω ότι αυτό πράγματι πρέπει να το συζητήσουμε και υπάρχουν αρκετέ περιπτώσεις που δείχνουν ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ε, ερωτώ λοιπόν, Ποιο πλήρωσε τελικά, οι κυβερνήσει, οι κατασκευαστέ, γιατί δεν υπάρχει ε, κάποια σαφή διαδικασία που να είναι μάλιστα εναρμονισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ερωτώ παρακαλώ, ε, έκανα αυτή την ερώτηση. Πολύ ωραία, η Έλενα. Και εγώ ε, θέλω να ρωτήσω σχετικά με τα κλινικά στοιχεία. Αναφερθήκατε στο ότι υπήρξε μια αλλαγή από το 2010. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε τι άλλαξε και γιατί ακριβώς το 2010. Εξάλλου πολλοί επέκριναν την κοινωνική νομοθεσία και λένε ότι το θέμα με τα κλινικά ε, δεδομένα στο Αμένο Βασίλειο είναι απλά μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Ε, δεν χρησιμοποιούνται ε, όπως ας πούμε στις Ηνωμένε Πολιτείε και διερωτώ με, μπορείτε να μου δώσετε κάποια απάντηση σε αυτό συγκεκριμένα. Το 2010 τι άλλαξε, διότι από ό,τι ξέρω στην περίπτωση των ισχύων άλλαξαν τα εξαρτήματα. Είναι ε, κομμάτια μέταλλο τα οποία επιπλέουν στο ανθρώπινο αίμα. Ε, υπήρχε παλαιότερα πρόβλημα, αυτό το έχει ομολογήσει τώρα ο κατασκευαστής, δηλαδή μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους στη δική μου την εκλογική περιφέρεια τουλάχιστον που ανησυχούν για τα επιτέματα αυτά, τα μεταλλικά ε, και πρέπει να υποστούν εξετάσεις αίματος. Βεβαίως ε, Όλοι λένε καλύτερα τα προϊόντα να βγαίνουν πιο γρήγορα στην αγορά. Αλλά το να βγαίνουν πιο γρήγορα στην αγορά δημιουργείται προβλήματα στους ασθενείς και δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Πολύ ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι. Ε, παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, για να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, ε, καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται, αλλά νομίζω ότι αυτό που ρωτήθηκε κατ' ουσίαν μπορεί να απαντηθεί από τα κράτη-μέλη. Εμπίπτει στη δική του συναρμοδιότητα, στην οργάνωση με την, τον τρόπο με τον οποίο έχουν οργανώσει τα συστήματα υγεία. Θα το ελέγξουμε, εν πάση περιπτώσει. Γνωρίζω, παραδείγματο χάρη, ότι ένα παρεμφερέ σύστημα υπάρχει και σε άλλου ε, τομεί, ε, παραδείγματο χάρη σε σχέση με της, ε, με ταξιδίων. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, πάντως μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό με τα κρατημέλη για να το μεταγίνει στο μέλλον, να υπάρχει κάποιος συντονισμός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο τέτοιου είδους ρυθμίσεις να τις εντάξουμε στην κοινοτική νομοθεσία. Όσον αφορά τώρα τα κλινικά δεδομένα. Το Έχουμε την οδηγία του 2007 2007 ναι. Και ε, λέει η οδηγία αυτή ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν κλινικές έρευνες. Δηλαδή, ο κατασκευαστής κατά κανόνα πρέπει να αποδείξει ότι έχει στη διάθεσή του κλινικά στοιχεία τα οποία απορρέουν μετά από μια έρευνα που είναι το αντίστοιχο της κλινικής δοκιμής για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Βεβαίως μπορούν να αποφύγουν αυτό μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν κάθε δικαίωμα να βασιστούν στα υπάρχοντα στοιχεία. Δηλαδή, αν το εξάρτημα αυτό μοιάζει με ένα άλλο που προϋπήρξε και για το οποίο υπάρχουν δεδομένα, τότε ναι. Όπως σας είπα λοιπόν, αυτά τα στοιχεία την εποχή που γινόταν αξιολόγηση πριν τοποθετηθεί το προϊόν στην αγορά, αντικαταστάθηκαν από ένα άλλο σύστημα ελέγχου. Και ο αρμόδιος φορέας που ενημερώνεται για αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να ενημερώνεται για προβλήματα που προκύπτουν που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επανεξέταση του εξαρτήματος. Όσον αφορά τώρα τα εμφυτεύματα ισχύου, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πράγματι δημιουργούνται προβλήματα με αυτά τα μεταλλικά εξαρτήματα τα οποία ενδέχεται να αποδεσμευτούν και να κυκλοφορούν στο αίμα του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτός λοιπόν είναι ένας κίνδυνος ο οποίος κατέστη σαφής μετά την ένταξη, τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Η, η, κυρία Μακεών, Μα αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει το πρόβλημα. Κατάλαβα ότι άλλαξαν τα εφητεύματα για το ισχύο ελαφρά. Και επειδή θεωρήθηκαν ισοδύναμα τα κλινικά στοιχεία, δεν χρειάστηκαν επιπλέον ε, ε, μελέτες και δοκιμές και μετά αρχίσαν να, βγαίνουν, να φεύγουν ρινίσματα από αυτά τα καινούργια για να μπαίνουν στο αίμα. Αυτό δείχνει ποιο είναι το πρόβλημα. Έχετε στοιχεία ε, ελέγχου και έρευνας της αγοράς, αλλά πρέπει ε, να ελέγξετε πώς λειτουργούν σε πραγματικά άτομα. Πώς αλλιώς θα ξέρετε τι έγινε. Χιλιάδες, πολλές χιλιάδες άτομα πήραν αυτό το καινούριο εφήτευμα χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτό πρέπει να εξετάσουμε ω ευρωβουλευτές. Υπάρχουν διάφορα τέτοια ε, ιατρικό-τεχνολογικά εξαρτήματα, αλλά τα βάζουμε στο σώμα μας. Και ορισμένα λέγεται ότι είναι και καρκινογενή. Είναι πολύ σοβαρό, ελπίζω λοιπόν η Επιτροπή να το ξαναδεί το θέμα. Βεβαίω η διαδικασία ακολουθήθηκε, αλλά ίσω δεν ήταν επαρκή η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μακιόν. Οπότε κλείνει η συζήτηση για το θέμα αυτό προθεσμία για υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 28 Μαρτίου. Στις 25 Απριλίου θα το συζητήσουμε, συγγνώμη θα το ψηφίσουμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην ε, πρώτη Ολομέλεια του Μαΐου θα υπάρξει η τελική ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, για τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Οπότε τώρα θα διακόψω τη συνεδρίαση μέχρι τις 11 και παρακαλώ όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ παρόντες να επανέλθουν με άλλους δύο ο καθένας ούτως ώστε όταν θα έλθουν συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουμε κι εμείς ε, αρκετούς παρόντες. Μισή ώρα λοιπόν διακοπή και ακριβώς στις 11 ξαναρχίζουμε. Ευχαριστώ.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 So, ich möchte... Please take... Παρακαλώ, καθίστε. Σας καλωσορίζω θερμότατα στην διακοινοβουλευτική συνεδρίαση για την προπαρασκευή της συνάντησης κορυφής Ρίο 20. Βλέπω ότι υπάρχουν αρκετοί παρόντες. Αυτό που θα γίνει στο Ρίο έχει ιστορικό χαρακτήρα, η ημερομηνία δηλαδή, και είμαι πεισμένος ότι και τα αποτελέσματα θα έχουν ιστορική σημασία, ότι η διάσκεψη αυτή στο Ρίο πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχει και θα επιτύχει. Θα επιτύχει εάν εμείς όλοι στην Ευρώπη, τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Επιτροπή, προετοιμάσουν καλά τη συνάντηση κορυφής, δείξουν περισσότερο το χαρακτήρα μας, θέσουν στην ημερήσια διάταξη αυτά τα θέματα που θέλουμε να υπάρξουν και κάνουμε σωστές διαπραγματεύσεις. Πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουμε σωστά. Και αυτός είναι ο στόχος της σημερινής συνάντησής μας με τους συναδέλφους από 20 χώρες και 23 κοινοβούλια. Και συνολικά Έχουμε 37 συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια παρόντες, προσκεκλημένους μας και από πλευράς της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Περιβάλλον. Σας καλωσορίζω στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και προσβλέπουμε στη συζήτηση που θα κάνουμε. Καλώς ορίσατε. Η συνεδρίαση σήμερα θα έχει δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα θέλουμε να συζητήσουμε πώς θα διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο για μια βιώσιμη περιβαλλοντική πολιτική και τι θα συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Και το δεύτερο τμήμα θα είναι μια συζήτηση για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης οικονομικής πολιτικής και μιας βιώσιμης ανάπτυξης που θα μας βοηθήσει να εξαλείψουμε τη φτώχεια αλλά να υπάρξει και βιωσιμότητα γενικότερα στους τομείς αυτούς. Και για το πρώτο τμήμα λοιπόν χαιρετίζω την ε, ομιλήτριά μας, την κύρια ομιλήτριά μας που είναι από τη χώρα που έχει αυτή τη στιγμή την Προεδρία του Συμβουλίου και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ε, Δανικού Κοινοβούλιου Φόλκετινγκ. Καλώς ήρθατε κυρία Λόκλιντ ε, στο Κοινοβούλιο και σας δίνω αμέσως το λόγο για την εισαγωγική ομιλία στην οποία όλοι προσβλέπουμε με μεγάλες προσδοκίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να σα απευθύνω το λόγο ω πρόεδρο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο ε, του ε, Δανικού ε, Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίση να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ κατάλληλη χρονική στιγμή για να συζητήσουμε το θέμα της προετοιμασίας του Ρίο 20. Έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θεσμικό πλαίσιο για την αηφόρο ανάπτυξη, ένα από τα βασικά στοιχεία του ε, σχεδίου υπαριθμών 0 για τα αποτελέσματα ε, που, τις διάσκεψεις που θα λάβουν χώρα στο ε, Ρίο Janeiro σε λιγότερους από τρεις μήνες. Αν δεν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις μας σίγουρα, σήμερα τουλάχιστον θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τη συζήτηση στη διακυβερνητική διάσκεψη στην Κοπενχάγη στις 14 και 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους, όπου οι τελικές προετοιμασίες για το Ρίο θα έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Πριν ε, συζητήσουμε το θέμα για, την, ε, για το θεσμικό πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ε, ένα αποτέλεσμα δράσης και προσανατολισμένου προς το μέλλον στο Ρίο. Θα είναι πολύ καταθλιπτικό και απογοητευτικό να συζητήσουμε απλώς τον απολογισμό από το 1992. Εγώ έχω τεράστιες προσδοκίες από τη διάσκεψη. Θα έπρεπε με το Ρίο Συν 20 να ε, ξεκινήσουμε μια προσπάθεια ε, μετάβασης προς την πράσινη ε, οικονομία, όπως επίσης και ε, να προετοιμάσουμε ένα ενισχυμένο θεσμικό πλαίσιο. Το έγγραφο αποτελεσμάτων θα πρέπει να στοχεύει, να είναι στοχευμένο, να είναι μια πολιτική δήλωση με ένα κοινό όραμα αλλαγής και μετάβασης, όπως επίσης και για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Πιστεύω λοιπόν ότι το εν λόγω έγγραφο ούτως ή άλλως το διαπραγματευόμαστε αυτές τις ημέρες και θα θέλα να δω, να συζητήσουμε τι ε, ζητημάτων μπορούμε να συζητήσουμε σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο αϊφόρου ε, αηφόρου ανάπτυξης, που είναι πάρα πολύ καθοριστικό για την επίτευξη των στόχων μας. Ε, αυτό Μπορεί να πει κάποιο ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από αυτό το έγγραφο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε για στόχου, ε, για δράσει, όμω ε, ε, τα επόμενα έτη είναι πάρα πολύ σημαντικά για την αηφόρο ανάπτυξη. Πρέπει εκτός από τις ε, συνδέσεις που έχουμε κάνει με την, ε, ε, με την φτώχεια, την μείωση των εθνικών πόρων και την υποβάθμιση του οικοσυστήματος, ο κατακαιρματισμός και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών είναι σύνηθες φαινόμενο. Πρέπει να σκεφτούμε ποιοι φορείς και οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών μπορούν να βοηθήσουν τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία σε ένα πλαίσιο αηφόρου ανάπτυξης και εξάλληψης της φτώχειας. Υπάρχει ένας ε, έτονος σύνδεσμος μεταξύ του θεσμικού πλαισίου και ε, άλλων ζητημάτων, όπως για παράδειγμα την πράσινη ανάπτυξη στο πλαίσιο της αηφόρου ανάπτυξης και της εξάλληψης της ε, φτώχειας. Εκτός από τους κανονισμούς, στους οποίους βέβαια πρέπει να σεβόμαστε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη συμμετοχής πολυμερών ε, οργανισμών και ιδρυμάτων. Ε, οι δομές ε, διακυβέρνησης είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικές για τι πράσινε οικονομίες και την εξάλληψη τη φτώχεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν ζητήσει μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου για την αηφόρο ανάπτυξη, για να μπορέσουμε να καλύψουμε, ε, να γεφυρώσουμε τα χάσματα και να επισπεύσουμε την παγκόσμια δράση. Αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση τη εφαρμογή των συμπεφωνημένων ε, ε, αποτελεσμάτων και των πρέπει να ενισχυθούν. Όπως αναφέρεται λοιπόν στο έγγραφο ε, αυτό, ε, πρέπει να σκεφτούμε το θέμα της αηφόρου ανάπτυξης. Ο τίτλος είναι πάρα πολύ καλός, αλλά και το μέλλον ε, πρέπει να αναφέρεται όλος ιδιαίτερος. Πρέπει λοιπόν πρώτα να ε, ενσωματωθεί η αηφόρος ανάπτυξη ως επιστέγασμα όλων των προσπαθειών ε, που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης πρέπει ενδεχομένως ε, να ε, αλλάξουμε την Επιτροπή ε, Αϊφόρου Ανάπτυξης σε Συμβούλιο Αϊφόρου Ανάπτυξης για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την Αϊφόρου Ανάπτυξη, την αποτελεσματική εφαρμογή σε όλα, το επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα όπως επίσης και την αποτελεσματική θεσμική συνοχή θα μας διευκολύνει στην συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, ε, ειδικότερα των μεγάλων ομάδων, ε, μέχρι εν ώψη της ε, διάσκεψης Ρίος 20. Υπάρχουν επίσης τρεις πτυχές παρακολούθησης και ρόλου που θα μπορούσε να ενισχύσει η ΕΚΟΣΟΚ όπως επίσης ε, και πολλά ζητήματα που πρέπει να διαπραγματευτούμε στο πλαίσιο της 67ης ε, Γενικής Συνέλευσης με τις υπόλοιπες ε, αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Η πτυχή της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης πρέπει να ενισχυθεί και εμείς εκφράζουμε την υποστήριξή μας για την, για αναβάθμιση του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, του UNEP είναι γεγονός ότι η ε, ε, η τρέχουσα κατάσταση διακυβέρνησης είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Κατά τις τα τελευταία 40 χρόνια έχουν ε, συναφθεί εκατοντάδες διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες και μάλιστα στο πλαίσιο 50 οργανισμών του ΟΗΕ για ποιο λόγο λοιπόν να μην υπάρξει ένα ειδικό, ένας ειδικός οργανισμός ε, βάσει του UNEP ε, που θα εδρεύει στο Ναϊρόμπι και το οποίο, ο θα μπορεί να ε, υποστηρίζεται από ένα σταθερό πλαίσιο επαρκών εισφορών για να μπορεί να βρίσκεται σε ισότιμη θέση με τους υπόλοιπους οργανισμούς του ΟΗΕ είναι γεγονός ότι πρέπει να αρχίσουμε με δράσεις στη δική μας χώρα. Το ε, Think Global Act Local, που ήταν ένα σύνθημα πριν από πολλά χρόνια, εξακολουθεί να ισχύει. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ενεργειακή πολιτική σε συνδυασμό με την αλληλευτική πολιτική, τη γεωργική πολιτική, την εμπορική πολιτική, την αναπτυξιακή πολιτική, την ε, οικονομική πολιτική, όλες τις πολιτικές ε, πρέπει να γίνει. Όλες αυτές οι πολιτικές πρέπει να συνεχίσουν συνάδουν με τους στόχους ε, της ε, της επίτευξης της αηφόρου ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, πρέπει να δούμε και τα ζητήματα τα ε, οικονομικά. η ισότητα είναι ένα σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο της αηφόρου ανάπτυξης. Στην αρχική δήλωση του Ρίο αναφερόταν και το θέλουμε και για το μέλλον και η κοινή και διαφοροποιημένη ευθύνη που πρέπει να έχουμε επίση αναφερόταν. Πρέπει να το λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο ε, ενθέρμο να εργαστεί προ την ενίσχυση τη τεχνολογία και τη τεχνογνωσία, ε, τη ανταλλαγή μάλιστα αυτών, για να ε, είναι τμήμα του Διεθνούς Μηχανισμού Διακυβέρνησης. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πτυχή ε, δεν διαχωρίζονται για να υπάρξει μια μοναδική ευκαιρία ε, συζητήσεων που θα στρέφονται προς το μέλλον ε, και που θα οδηγούν στην καλύτερη εφαρμογή και ε, την καλύτερη ενσωμάτωση της ε, πτυχής αηφόρου ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις χώρες. πώς μπορούμε, πώς μπορούμε όμως να διευκολύνουμε φιλόδοξο αποτέλεσμα στο Ρίο. Είναι γεγονός ότι η, η κατάσταση μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο σύγχρονη έννοια της ανάπτυξης και της χρήσης των πόρων μας που όλων Λοιπόν, όλο και λιγοστεύουν. Η, ε, η, αξιοποίηση, αξιοποίηση των πόρων είναι ένα βασικό στοιχείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοστάτη στην προσπάθεια αυτή. Το ε, να ε, συμμετέχουμε σε μια κοινή θέση για έναν πράσινο ε, χάρτη πορείας στο πλαίσιο του ΟΗΕ είναι κάτι που θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα και έχει άμεση σχέση με τα ζητήματα που έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και που θα συζητήσουμε ακόμη φέτος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά την άποψή μου, πρέπει να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε πριν από την ε, διάσκεψη την ευρωπαϊκή θέση, γιατί είναι μια μοναδική δυνατότητα για την παγκόσμια κοινότητα να, κάνει φιλόδοξες, ε, να αναλάβει φιλόδοξες δεσμεύσεις για ζητήματα περιβαλλοντικά. Και νομίζω ότι θα έπρεπε ως βουλευτές να συμμετέχουμε και να διευκολύνουμε τα αποτελέσματα με διάφορες διόδους. Και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ε, στην διάσκεψη της Globe International ε, που είναι μια οργάνωση βουλευτών με ε, σκοπό δημιουργίας κρίσιμης μάζας νομοθεσίας που σκοπό έχει να αντιμετωπίσει, να εξετάσει νομοθετικές απαντήσεις σε διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα. Από τις 15 ως τις 17 Μαΐου θα λάβει χώρα, συγγνώμη Ιουνίου, πριν από την διάσκεψη. Είμαι σίγουρη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει ενεργό λόγο στο πλαίσιο της διάσκεψης αλλά και πριν από αυτήν. Πρέπει να ε, δημιουργήσουμε γέφυρες συνεργασία με του εταίρου μας σε όλο τον κόσμο και ε, όλοι έχουν ένα ρόλο να διαρματίσουν. Ε, θα ήθελα να υπολογίζω στην βοήθειά σας και σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Λόνι Λόκλεντ για την ομιλία σας, τη βασική ομιλία. Οπότε τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναφερθώ στη διαδικασία για τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε πάνω στο τραπέζι ε, χαρτιά σας παρακαλούμε λοιπόν να ε, σημειώσετε ότι θέλετε να γράψετε, να σημειώσετε ότι θέλετε να μιλήσετε σε αυτά τα χαρτιά της κάρτες ε, ε, και θα τα συγκεντρώσουμε. Οι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρουν πώς δίνουμε το λόγο και από πλευράς ε, διαδικασίες θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο, να δίνουμε το λόγο σε δύο συναδέλφου από Εθνικά Κοινοβούλια και μετά σε έναν συνάδελφο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ όλου του συναδέλφου να τηρήσουν ένα χρόνο δύο λεπτών, ούτω ώστε να μπορέσουν να πάρουν το λόγο όλοι οι συνάδελφοι που το επιθυμούν. Δεν έχουμε μόνο συναδέλφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια εδώ, αλλά και από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι ο κύριο ε, Στέφαν Νίλσον παρόν, γιατί και αυτό το θεσμικό όργανο ασχολείται έντονα με την προετοιμασία του Ρίο και φυσικά έχουμε την Επιτροπή Περιφερειών. Ο Μισελ Λεπούν είναι ο εκπρόσωπος εδώ στο Προεδρείο και φυσικά ε, και εκείνο θα να καλωσορίσω. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Αδάμου από την Κύπρο, τον οποίο καλωσορίζω εδώ στο Κοινοβούλιο. Στον κύριο Αδάμου λοιπόν το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Χαίρομαι που επανέρχομαι έστω και με την ιδιότητα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή τη Βουλή των Αντιπροσώπων τη Κύπρου. Έχω θητεύσει εδώ πέντε χρόνια. Χαρά που σα βλέπω ξανά όλου. Αναφίβολα η πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα τη αηφόρου ανάπτυξη στα 20 σχεδόν χρόνια που έχουν παρέλθει από την ιστορική διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που έλαβε χώρα στο Ρίο το 1992, είναι σημαντική. Οι νέε όμω προκλήσει που προκύπτουν από τι άμεσε επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή και τη οικονομική εξαθλίωση την οποία έχουν οδηγηθεί οι συνάνθρωποι μα από το παγκόσμιο, λόγω φυσικά τη οικονομική κρίση που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία απαιτούν τη λήψη άμεση δράση στο διεθνέ και εθνικό επίπεδο για την προώθηση τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα πρέπει να έχει ω επίκεντρο τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι η πιο δόκιμη μέθοδο ενδυνάμωση του περιβαλλοντικού προγράμματο των Ηνωμένων είναι αυτή που έχει άλλωστε εισηγηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή με την πιθανή μετατροπή του σε εξειδικευμένο οργανισμό που να λειτουργεί εντό του συστήματο των Ηνωμένων στη βάση του προτύπου άλλων οργανισμών των ΗΕ Εθνών, για παράδειγμα το ILO ή το FAO. Η αποτελεσματικότητα του εν λόγω οργανισμού θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με τη δημιουργία επιστημονική επιτροπή για τεχνοκρατική στήριξη του έργου του, αλλά επίση και με την παροχή τη απαραίτητη αρμοδιότητα για τη διαχείριση των θεμάτων που θα αφορούν την αεφόρο ανάπτυξη έτσι ώστε να αποφευθεί η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που οδηγεί σε σύγχυση αλλά και καθυστέρηση στην ανάληψη δράση. Τελειώνοντα, ευελπιστώ ότι το σχέδιο δράση για το περιβάλλον και την αηφόρο ανάπτυξη, το οποίο θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του 2012, θα ανανεώσει την πολιτική δέσμευση τη Ένωση για την αηφόρο ανάπτυξη, η οποία να αντιμετωπίζει τι υφιστάμενε αλλά και τι νέε προκλήσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, ο συνάδελφος Απαρίθη. Δεν ξέρω πού είναι. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Απαρίθινο είναι το όνομά μου. Σχεδόν τέλεια το προφέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Παίρνω το λόγο, καταρχάς, ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι ως ε, ε, γερουσία της Ισπανίας που είμαστε εδώ μαζί με πολλούς άλλους ε, βουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από άλλες χώρες. Πιστεύουμε ότι είναι θαυμάσια ιδέα αυτή η συνεδρίαση. Χαιρετίζουμε λοιπόν με θετικό και σαφή τρόπο αυτή τη συνεδρίαση. Θεωρούμε ότι το Ρίο Συνήκος είναι μια νέα ευκαιρία, μια νέα σημαντική ευκαιρία, ούτω ώστε να οδεύσουμε όλοι μαζί προς μια πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη. Θα θέλαμε να είναι πολύ πιο επιτυχημένη αυτή η συνεδρίαση σε σχέση με την προηγούμενη πριν από 20 χρόνια όλες οι διαδικασίες που ξεκίνησαν σε αυτή την προηγούμενη με στόχο μια βιώσιμη ανάπτυξη όπως πραγματικά την εννοούμε όλα αυτά δεν είχαν την επιτυχία που όλοι αναμέναμε. Γι' αυτό επιθυμούμε τώρα και γι' αυτό είμαστε εδώ να υπάρξει ενότητα όλων των χωρών ούτω ώστε να επιτύχουμε την εκπλήρωση αυτών των στόχων που μας ε, παρουσίασε και η συνάδελφος από την Δανία, με την οποία συμφωνούμε απόλυτα. Θέλουμε να εργαστούμε μαζί ως γερουσία της Ισπανίας για να προωθήσουμε αυτούς τους στόχους που έχει θέσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όποτε μας χρειαστείτε θα ερχόμαστε για να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. ο συνάδελφο Γκαμπράντη, που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, του Κοινοβουλίου που θα πάει στο Ρίο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ματία. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ τη Λόνα για την ε, συμμετοχή της. Ε, κλείνουμε τις ε, κουρτίνες, τα στόρια, οπότε μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. πολύ περισσότερο από πριν. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υποτιμήσουμε το ρόλο μας ως ευρωβουλευτών. Πιστεύουμε ότι για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό τμήμα του να είμαστε εδώ και εσείς ως εθνικοί βουλευτές και εμείς ως ευρωβουλευτές. Πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας να είναι πιο φιλόδοξες ε, εν ώψη του Ρίο 20. Η Σύνοδος Κορυφής του 1992 έδωσε ε, στην περιβαλλοντική σκέψη μια τεράστια όθηση. Ορισμένοι ξέρω, πως είπαν, ότι δεν ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα, αλλά δεν θα έπρεπε να υποτιμούμε το τι ε, συνέβη στο μυαλό πολλών ανθρώπων χάρη στο 1992 και ε, πραγματικά πιστεύω ότι η διάσκεψη ε, του Ιουνίου φέτος ε, θα μπορέσει να κάνει το ίδιο. Για μένα το σημαντικό, εκεί που καταλήγουμε δηλαδή, είναι η καλή διαχείριση των, των ε, φυσικών πόρων. Όλο περισσότερο φτάνουμε στα όρια της ε, των πόρων αυτών και είναι κάτι το οποίο έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του ε, Ρίο ε, ε, Πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν το κλιματικό περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή είναι πολύ σημαντικά. Σε πολλές περιπτώσεις ολόκληρη οι κλάδοι έχουν παραλύσει σε μερικές χώρες μέλη. Είναι πραγματικά περίεργο το διεθνές ε, ελεύθερο εμπόριο να είναι, όλο και περισσότερο σημαντικό στο πλανήτη μας. Έχουμε τον ΠΟΕ που δίνει τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών, αλλά αυτό που λείπει είναι κάτι τέτοιο σε επίπεδο ε, περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών ζητημάτων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα ε, σημαντικό στοιχείο του Ρίο Συνήκωση, να μπορέσει σε διεθνές επίπεδο να οργανώσει ένα πολύ ισχυρότερο φορέα του ΟΗΕ σε σχέση με αυτόν που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρω δύο λεπτά έχω στη διάθεσή μου, ε, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό θα ολοκληρώσω. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε ένα διεθνή φορέα τύπου ΠΟΕ για το περιβάλλον. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι θα μας επέτρεπε να προοδεύσουμε ε, ακόμη περισσότερο. Θα ήταν καλύτερο να έχουμε, όπως λέμε και στο ψήφισμά μας, ε, ένα διεθνές δικαστήριο για το περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι ε, προτεραιότητα στο, στην ημερήσια διάταξη των κυβερνήσεων για το Ρίο. Να δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρο της οικονομικής, στον πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τον Στέφαν Νίλσον. Και πάλι σας καλωσορίζω, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα να σας μιλήσω από την κοινωνία των πολιτών. Είμαστε το μόνο σώμα που αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Απαιτούμε η συνδιάσκεψη να δεσμεύσει τους ε, ηγέτες όλων των κρατών να εξαλείψουν την φτώχεια, να προστατεύσουν τον πλανήτη, να προωθήσουν μια πράσινη οικονομία. Όλα αυτά είναι τμήματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών, οικολογικών και οικονομικών πλευρών της ανάπτυξης. Υποστηρίζουμε λοιπόν, τα λέω επιγραμματικά, η Επιτροπή Αϊφόρου Ανάπτυξη να αντικατασταθεί με ένα Συμβούλιο Αϊφόρου ανάπτυξη, με ένα σύντομο, ισχυρό, σύντομη ισχυρή εντολή. Πιστεύουμε επίσης ότι το πρόγραμμα των ΗΠΑ θα μπορούσε να γίνει ένα νέο φορέα για το περιβάλλον, με καλύτερη και ισχυρότερη εντολή. Και θέλουμε και η κοινωνία των πολιτών να εμπλακεί σε όλες τις κύριες προσπάθειες και ομάδες και συζητήσεις στο μέλλον. Επίσης θα θέλαμε ο Ombudsman για τις επόμενες γενιές να υπάρξει ο στασμός. Επίσης υποστηρίζουμε την πρόσβαση της κοινή γνώμης στην πληροφόρηση για τα θέματα αυτά. Και ακόμη, το Συμβούλιο να δώσει εντολή, και εδώ έχετε μεγάλο ρόλο να παίξετε, να στηρίξετε το Συμβούλιο, να δώσει εντολή στην Επιτροπή να μπορεί να είναι εκπρόσωπός μας, να διαπραγματεύεται με μια φωνή. Αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να επιτύχει αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα αυτή σε δύο λεπτά να περιγράψω αυτά που θέλω να πω. Με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος, που είναι περιορισμένος ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, Περιφερειών Φεθαλαστολών, κ. Λέπνη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα στην Επιτροπή Περιφερειών ε, να τοποθετηθεί. Η πρόεδρός μας, η κυρία Μπρεζό, δυστυχώς έχει ελλημένες υποχρεώσεις και δεν μπορεί να παρίσταται. Αυτό που ζητάει η Επιτροπή Περιφερειών είναι βεβαίως ε, να προσυπογράψει ε, μία ε, στρατηγική διακυβέρνηση σε πολλών επιπέδων με αλληλεπίδραση, με συνέργειες και συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των επιπέδων εξουσίας. Επομένως, στο πρώτο αυτό σχέδιο του τελικού εγγράφου χαιρόμαστε που υπάρχουν θετικές αναφορές σε σχέση με το ρόλο των τοπικών αρχών. Βλέπω ότι αναφέρεται στο κείμενο, όμως μου φαίνεται ότι τέσσερις άξονες χρειάζονται για να το συμπληρώσουν. Πρώτον, θα θέλαμε μια ενισχυμένη διακυβέρνηση σε διεθνές επίπεδο με την ε, μεταρρύθμιση του προγράμματος ε, του ΟΗΕ για το περιβάλλον σε πραγματικό οργανισμό και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Γερμπράντη σχετικά. Δεύτερον, ζητούμε οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, να αναγνωρίζονται ε, στο θεσμικό πλαίσιο ε, όπως και οι εθνικές κυβερνήσεις και ε, οι φορείς του ΟΗΕ ως κυβερνητική ε, εταίροι πλήρω αναγνωρισμένοι. Επίση, πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη διακυβέρνηση σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μετά από τη ε, διάσκεψη του Ρίο του 1992 ε, σε διάφορε υπήρου και στην Ευρώπη μάλιστα. Άρχισαν να ισχύουν οι τοπικέ αρχέ, να εμφανίζονται τοπικέ αρχέ και εμεί θα θέλαμε να αναβιώσει αυτή η προσπάθεια που άρχισε το 1992. Τρίτον, ζητούμε, όπω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ρίο Συνήκωση να υποστηρίξει την περιβαλλοντική δημοκρατία σε διεθνές ε, επίπεδο, υποστηρίζοντας, ε, για παράδειγμα, ε, άλλες συμβάσεις περιφερειακού χαρακτήρα, παρόμοιες με την σύμβαση του Άρους και τέταρτο στοιχείο, θα ολοκληρώσω έτσι, το θεσμικό πλαίσιο της αηφόρου ανάπτυξης που θα αποφασιστεί στο Ρίο πρέπει να συμπεριλάβει ένα χάρτη πορείας για ε, την ε, ε, ύπαρξη στόχων στο πλαίσιο της αηφόρου ανάπτυξης με πολύ συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες πρέπει να προβούμε και συγκεκριμένα μετρήσιμα εργαλεία για να είναι μετρήσιμοι και οι στόχοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συμβολή σας. Και τώρα ζήτησε το λόγο ο συνάδελφος Μπρίνκερτ από την Μάλτα. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το καυτό θέμα της ε, ανάπτυξης και συμφωνίες επί των ε, στόχων αεφόρου ανάπτυξης πρέπει να είναι αντικείμενο συμφωνίες και καλής διάρθρωσης. Ιδιαίτερα επειδή οι στόχοι για την ανάπτυξη της ε, χιλιετίας δεν έδωσαν αρκετή σημασία στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Αλλά πριν ορίσουμε ποιοι είναι οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι, τουλάχιστον να έχουμε την πολιτική δέσμευση για το αν πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι στόχοι ή όχι. Κάποιος πρόσφατα είπε ότι η πολιτική δεν πρέπει να ασχολείται με την βιώσιμη ανάπτυξη. Χωρίς πολιτική όμως δεν θα κερδίσουμε την καρδιά και το μυαλό, δεν θα επιτύχουμε τον σφαιρικό αυτό στόχο. Γι' αυτό πιστεύω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, κυβερνήσεις, βουλευτές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, όλοι οι άλλοι φορείς και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να επιδιώξουν σαφήνεια και συγκεκριμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, θεωρώ ότι και σε επίπεδο θεσμών και οργανώσεων των ΗΕ πρέπει να ενισχυθεί η ίδια υποδομή που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Βεβαίως πρέπει να προετοιμάσουμε σωστά το επερχόμενο Ρίο συνήκωση. Πρέπει ήδη να δούμε πώς θα προετοιμάσουμε και την περίοδο μετά το Ρίο. Ήδη τώρα να προετοιμάσουμε στόχους, προθεσμίες και πολύ σαφή κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπρίνκατ, επόμενος. Ο κύριος Ιτάλγο από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. από πλευρά τη ισπανική Γερουσίας και των Ισπανών Σοσιαλιστών θέλω να ανακοινώσω τη δέσμευσή μας συμφωνώντας με όλες τι προτάσεις και ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των διαφόρων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πάνω απ' όλα με την ε, έκθεση υψηλού επίπεδου των Ηνωμένων Εθνών για την ε, παγκόσμια βιωσιμότητα στην οποία συμμετείχε η σύντροφός μας και Υπουργός Περιβάλλοντος Χριστίνα Ναρμόνα. Οι προτάσεις και συστάσεις είναι πιο αναγκαίες παρά ποτέ αυτή τη στιγμή που υπάρχει οικονομική κρίση παγκοσμίω. Η κρίση αυτή προκλήθηκε από την χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να επιληφθεί. Αλλά είναι και ευθύνη του καθενός μας για αντιμετώπιση τη κρίση με βάση το επίπεδο υπευθυνότητα που μπορούμε να έχουμε σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Υποστηρίζουμε όλε τι προτάσει, ούτω ώστε να υπάρξει μια θεσμική δομή σε παγκόσμιο επίπεδο με νέου οργανισμού, νέε ομάδε εργασία για να υπάρξουν συμμαχίε. Μια σφαιρική δράση σε όλα τα επίπεδα κυβέρνηση. Να υπάρχουν μηχανισμοί επιστημονική βοήθεια, ρυθμιστικοί μηχανισμοί και να λειτουργούν σε τοπικό, κρατικό και παγκόσμιο επίπεδο. Όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε να αλλάξει η στη διάταξη λόγω τη ε, παγκόσμιας κρίσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η κρίση δεν μπορεί να είναι η δικαιολογία για να μειώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, για να μειώσουμε τι προσπάθειε να διατηρήσουμε καθαρές τι ακτές μα. Η κρίση δεν πρέπει να είναι το πρόσχημα για να μην συνεχίσουμε να βοηθάμε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Η κρίση δεν πρέπει να καταργήσει ούτε τη βιωσιμότητα, ούτε το περιβάλλον, τα δικαιώματα των εργαζομένων γιατί παίζεται το μέλλον του πλανήτη μας και το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι σε αυτό το πλανήτη ζούμε. Όλα τα μέσα αυτά λοιπόν και τα μέτρα είναι επίγοντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ιδάλγο. Ρίχαρτ Πρόεδρε, θέλω να υπενθυμίσω ότι αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα των υδάτων και επίση ότι επιτύχαμε τον πρώτο στόχο τη χιλιετία που είναι η πρόσβαση σε καθαρό ε, πόσιμο νερό για 98% των πολιτών του κόσμου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εξελίξει ε, που πρέπει να αναφερθούν. Το νερό βεβαίω και βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαρτιών μα ε, αν θέλουμε να επιτύχουμε και του υπόλοιπου στόχου τη χιλιετία. Έχουμε περίπου 9,3 δισεκατομμύρια ανθρώπου γή περίπου ε, κατά 70% έχει αυξηθεί η ζήτηση για τρόφιμα και παρατηρείται και έντονη αστιφιλία. Συγκεντρώνονται οι άνθρωποι σε αστικά κέντρα. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες η γεωργία τόσο όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων όσο και όσον αφορά το γεωργικό εισόδημα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου κυρίως τη μικρή γεωργία, αυτή να προβάλλουμε έχοντας ε, κυρίως ε, κατά νου ότι με τον τρόπο αυτό ε, στηρίζουμε τις γυναίκες γιατί οι γυναίκες είναι κατά, λόγο, κατά κύριο λόγο υπεύθυνε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εστιάσει την προσοχή της στη συνεργασία στα κρατημέλη, να εστιάσει την προσοχή της σε κέντρα ε, αστικής συγκέντρωση. Ε, σας υπενθυμίζω τα προβλήματα που υπάρχουν στο Κασμίρι, στην Ινδία, στο Πακιστάν. Τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να ασχοληθούν με τις περιπτώσεις αυτές έτσι ώστε να στηρίξουν και να προβάλλουν την ειρήνη. Εξάλλου, οφείλουμε να έχουμε σωστή χρηματοδότηση κυρίως για τις στατικές υποδομές, για την άρτευση-ίδρυυση. Ε, αναφέρομαι γενικότερα στο νερό. Στον τομέα της γεωργίας θέλω επίσης να επενθυμίσω ότι πρέπει να προβάλλουμε προσιτές τιμές τεχνικές ε, υδροδότησης. Ε, νομίζω ότι το οφείλουμε αυτό στους εταίρους μας ε, στα κράτη-μέλη. Γιατί αν δεν προβάλλουμε το νερό στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους υπόλοιπους στόχους της ε, χιλίτιας. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος ε, και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Χάιντεχριχ από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ονομάζομαι Χέλμουτ Χάιντεχριχ. Εγώ είμαι μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία και είμαι ευγνώμων που μας δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να έρθουμε εδώ ως βουλευτές των Εθνικών και να συζητήσουμε μεταξύ μα. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η συζήτηση για την εξέλιξη του κλίματος ε, στην Ευρώπη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, κυρίως σε αυτήν την εποχή κατά την οποία προσπαθούμε να ε, μεταβούμε σε μια νέα μορφή ενεργειακού εφοδιασμού στη Γερμανία και με νέες μορφές να εφοδιάζουμε με ενέργεια το σύνολο της Γερμανίας. Ελπίζω λοιπόν ότι στις ε, διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις δεν θα συζητήσουμε γενικά για στόχους, αλλά πολύ συγκεκριμένα για συγκεκριμένες συμφωνίες να συνομολογήσουμε συμφωνίες, να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Θέλω λοιπόν να πω ότι κατά την άποψή μας οι εξελίξεις ε, θα στεφτούν από επιτυχία μόνο εφόσον ε, τα κράτη-μέλη αναλάβουν υποχρώσεις ε, που θα μπορούν να ελεγχθούν ως προς την υλοποίησή τους, μόνο αν έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Μόνο εάν τα κράτη-μέλη στην πράξη σημειώσουν πρόοδο και γενικότερα ε, προοδεύσουν στην ε, ανάπτυξη, όσον αφορά στην ανάπτυξη. Ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω, γιατί ο προαλής σας μίλησε για το νερό. Εμείς λοιπόν στηρίζουμε την διασύνδεση της ανάπτυξης με την ενέργεια. Ακριβώς αυτό που είπε προηγουμένως και η προλαλήσασα, ε, που μίλησε για τη διασύνδεση γεωργίας και διαχείριση νερού. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι εγώ έχω καταθέσει συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να προβληθεί περισσότερο το θέμα των υδάτων. Τελειώνοντας λοιπόν, θέλω να πω, εμείς ελπίζουμε ε, στα αποτελέσματα της συνδιάσκεψης του Ρίο να ενταχθούν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στο να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την εξέλιξη του παγκόσμιου κλίματος. Ευχαριστούμε και εμείς, λέει ο Πρόεδρος, και από τη Γαλλική Γερουσία έχει το λόγο η συνάλληση κυρία Ροσκινιόλ. Καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ευχαριστήσω ε, όσοι οργάνωσαν ε, αυτήν την συνάντηση. Μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε μαζί εθνικοί βουλευτές και ευρωβουλευτές. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική εργασία της όσον αφορά την πρότασή της. Για μας είναι μια βάση εργασίας πάρα πολύ σημαντική και πολύ φιλόδοξη. Επίσης, αναφέρει πάρα πολλές από τις ανησυχίες μας ε, εν ώψη του Ρίο Συνήκωση, για παράδειγμα ε, το θέμα της ε, της κοινή γνώμης η οποία αδιαφορεί για το θέμα αυτό όπως επίσης και το θέμα της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών. Νομίζουμε ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν σημαντικό ρόλο να διαγραμματίσουν ε, για την κοινοτοποίηση των, ε, της κοινή γνώμη, ε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχουμε τίποτα αν δεν συμμετέχει η κοινή γνώμη. Και αν τα εθνικά κοινοβούλια δεν ε, δεσμευτούν, ε, δεν επενδύσουν στην προετοιμασία, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Πρέπει να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή προσπάθεια και νομίζω ότι στο Ρίο Συν 20 μπορούμε να έχουμε την ίδια Ευρώπη που είχαμε και στον Τιρμπάν, φιλόδοξη και ενωμένη, γιατί ε, σήμερα είμαστε εδώ βουλευτές ειδικοί για τα θέματα τα περιβαλλοντικά. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας για τις δυσκολίες. Εξέρουμε τα προβλήματα, είτε είμαστε φιλελεύθεροι ελεύθεροι, είτε είμαστε δεξιοί, είτε είμαστε σοσιαλιστές, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, γνωρίζουμε Ποια είναι αυτά και χρειαζόμαστε όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να πείσουμε όσους κάνουν πολιτική μαζί μας για να ε, μην υπάρχουν τόσα πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα και να ξεφύγουμε από όλες αυτές τις περιβαλλοντικές απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και η σημερινή συνεδρίαση συνηφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση. Κύριος Γιολάνεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να είναι το βασικότερο θέμα κατά τον 21ο αιώνα. Ακούσαμε λοιπόν ότι είμαστε 9 ή 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη γη και καταλαβαίνετε εδώ ελοχεύει κίνδυνος ο απολογισμός από την πρώτη συνδιάσκευτο μέχρι σήμερα δεν είναι ικανοποιητικός. Το χάσμα ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους διευρύνθηκε. Στην οικονομία έχουμε την ε, στρέβλωση της ε, χρηματοδοτικής πολιτικής και της πραγματικής πολιτικής και το αποτύπωμα του άνθρακα ούτε και αυτό βελτιώθηκε. Νομίζω λοιπόν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα καθοριστική σημασία ε, θέμα και ελπίζω στο Ρίο να προκύψουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, στόχοι, χρονοδιαγράμματα και να τηρηθούν από όλου. Όπω και πολλοί άλλοι, και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλου. Δεν μπορούν να υλοποιήσουν όλα αυτά μόνε του οι κυβερνήσει. Χρειαζόμαστε τα κοινοβούλια, την τοπική αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών. Άρα δηλαδή είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλου. Και πρέπει να συζητηθεί ανοιχτά το τι μπορεί να κάνει να προσφέρει ο καθένα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαράξει μια στρατηγική βιώσιμότητα, αλλά δεν έχει προχωρήσει αυτό. Και συμφωνώ με τη συνάδελφο από τη Γαλλική Γερουσία ότι πράγματι χρειαζόμαστε στρατηγικές ε, βιώσιμης ανάπτυξης από τη βάση μέχρι την κορυφή. Και εάν ε, στο Ρίο συζητήσουμε για την κορυφή, δηλαδή για, την, ε, για το παγκόσμιο επίπεδο αυτής της πολιτικής, τότε θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να μετατραπεί σε ένα είδος οργανισμού, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να επιβληθεί ο οργανισμός αυτός στους άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Πέρα από αυτό χρειαζόμαστε και ένα συμβούλιο βιωσιμότητας, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Δηλαδή ένα συμβούλιο, έναν οργανισμό, ο οποίος θα ελέγχει την εφαρμογή των συμφωνιών, ε, θα πρικοδοτηθεί με αρμοδιότητες για να υποβάλει και άλλες ερωτήσεις, ενδεχομένως και να υποβάλει, επιβάλλει και κυρώσεις. Αλλά κατά κύριο λόγο θα καταθέτει εκθέσεις, θα ελέγχει το κατά πόσον υλοποιούνται οι υποχρώσεις, όχι μόνο δηλαδή να προβαίνουμε σε ευχολόγια προθέσεις δηλώσεων και στην πράξη να μην συμβαίνει τίποτα. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να προβάλλουμε την Ευρώπη. Στο Ρίο καλούμεθα να αναλάβουμε ηγετική θέση. Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Τώρα Δίνω το λόγο στον πρόεδρο της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος από το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ε, διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης που μας επιτρέπει να ενημερωθούμε για τις απόψεις ημέν των ΔΕ. η παρουσίαση της εκπροσώπου του Συμβουλίου της Δανέζικης Προεδρίας μας είπε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μια σειρά από θέματα. Από αυτά εγώ θέλω να τονίσω ότι φέτος ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από την πρώτη συνάντηση και επίσης έχουμε και την έκθεση Μπρούντλαντ που είχε γίνει τότε. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κοινή μα θέση, όπω ακριβώ την παρουσίασε η εκπρόσωπο τη ε, δανέζικη κυβέρνηση, τονίζει ότι πρέπει η Ευρώπη να έχει επαφέ με όλε τι άλλε περιοχέ του κόσμου, με τη Βραζιλία, την Ιδία, την Κίνα. Δεν μπορούμε να είμαστε απομονωμένοι, γιατί θέλουμε ένα παγκόσμιο αποτέλεσμα. Μόνο ένα τέτοιο παγκόσμιο αποτέλεσμα θα είναι αποτελεσματικό. Αλλιώς η θέση μας ε, δεν θα μπορεί να έχει τον αντίκτυπο που θα έπρεπε να έχει. Αυτό νομίζω πως είναι το βασικό θέμα. Και δεύτερον, για την ίδια την κοινή μας θέση, να μην επαναλάβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα σφάλματα που δεν θα προωθήσουν μια ευφυή, πράσινη οικονομία που θα, μας που θα συμπεριλαμβάνει όλους. Γιατί υπήρξαν ε, σφάλματα κατά την ε, εκπόνηση της στρατηγικής της Λισαβόνας αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το 2020 και για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, χρειαζόμαστε μια σφαιρική προοπτική να δεσμευτούμε αποφασιστικά για να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας τα προβλήματα. Πρέπει να είναι δεσμευτική η νέα σύμβαση. Δεν θα την επιτύχουμε βέβαια στο Ρίο, αλλά τουλάχιστον να διευκρινίσουμε τους στόχους. Να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης που να προκύψει από αυτή τη συνάντηση κορυφής. Αυτή θα ήταν η έκκληση που θα ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα στον, ε, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ε, Βελικής Βουλής, την κυρία Νουά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ε, συνάδελφοι. Είμαι εδώ σαν αντιπρόεδρος ε, του ε, Υπουργείου του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι εδώ ο συνάδελφος γιατί έπρεπε να παραστεί στην κηδεία των παιδιών που ήταν θύματα του δυστυχήματος στην Ελβετία. Ε, θα ήθελα να σας πω ε, τι ζητούμε εμείς από την βελγική κυβέρνηση αλλά και ε, από όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας τι θέλουμε να υπερασπιστούν στην διάσκεψη του Ρίο και θα ήθελα να τονίσω ορισμένε πτυχές όσον αφορά την διακυβέρνηση. Στο ψήφισμα ως προς την διακυβέρνηση επιμείναμε σε δύο σημεία ε, την ενίσχυση δηλαδή του προγράμματος του ΟΗΕ για το περιβάλλον ε, με, δημιουργώντας έναν φορέα αντί για ένα απλό πρόγραμμα ε, και Πιστεύουμε ότι στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης είναι σημαντικό να δώσουμε μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό το πρόγραμμα ε, και μπορούμε έτσι να δώσουμε και μεγαλύτερη δύναμη και σε άλλες πολυμερείς ε, συμφωνίες ε, για το εμπόριο για παράδειγμα. Οπότε θα θέλαμε να αναφέρετε ότι οι συμμετέχοντες στη, διασκευή, στη διάσκεψη πρέπει να προβούν σε στρατηγική που να εξασφαλίζει τη συνοχή των διαφόρων πολυμερών συμφωνιών και μία συντονισμένη δράση για την απερίμωση, για την βιοπικιλότητα ε, και για την αηφόρο ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι αυτά τα σημεία πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε. Δεύτερη πτυχή ε, είναι οι δείκτες. Να μπορούμε δηλαδή να μετρούμε την πρόοδο που έχουμε κάνει ή που δεν έχουμε κάνει και να μπορέσουμε επίσης ε, να δουλεύουμε επί τη βάση ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης. Το Ρίο πρέπει να δώσει τη δυνατότητα μιας ε, εναλλακτικής μεθόδου ε, ευημερία ε, και ανάπτυξης και όχι μόνο να αναφερόμαστε σε δείκτες που βασίζονται στο ΑΕΠ. Ε, υπάρχουν, πρέπει να έχουμε δείκτες ε, ανθρώπινης ανάπτυξης. Ε, το πρόγραμμα του ΟΣΑ που αφορά την ανάπτυξη στο πλαίσιο της κοινωνίας και την ένταξη την κοινωνική και νομίζουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι σφαιρικά, συμπεριλαμβάνουν δηλαδή πολλές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ε, οικονομικές πτυχές. Αυτοί οι δείκτες θα μας δώσουν τη δυνατότητα χρήσης ενός μοντέλου πολύ πιο περιεκτικού ε, που ε, σέβεται τα όρια της, των οικοσυστημάτων. Για την πράσινη οικονομία θα τοποθετηθώ το απόγευμα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ούτσκι. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω όλους τους αδέλους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει μεγάλη σημασία. Αναμφίβολα. Να αντιδράσω στην ομιλία της κυρίας Λόκλιντ. Την εισαγωγική ομιλία λοιπόν. Πιστεύω ότι χρειάζονται θεσμικές αλλαγές, αλλά ίσως χαθούμε τελικά σε αυτές. Σε τελευταία ανάλυση οι εθνικές κυβερνήσεις λαμβάνουν τις αποφάσεις και επαναλαμβάνω ότι χωρίς σφαιρική συμφωνία με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Φοβάμαι ότι στις προσπάθειες να διαμορφώσουμε το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να χάσουμε το στόχο από τα μάτια μας. Θα πρότεινα λοιπόν να μην είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι στους στόχους μας, γιατί δεν επιτυχάνουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Ένα αποτέλεσμα που ανέφερε ο κύριος Ζήμπερ είναι η ίδρευση. Και εγώ συμμερίζομαι την άποψή του για τη σημασία του πόσιμου νερού, ας είναι αυτό ένα σημαντικό θέμα στο Ρίο Συνήκωση. Επίσης η διαχείριση των αποβλήτων. Και εδώ ο πλούσιος βοράς μπορεί να βοηθήσει τον ε, φτωχό νότο όπου υπάρχει πρόβλημα με την ε, διαχείριση των υδάτων. Ας επιδιώξουμε λοιπόν μικρά συγκεκριμένα βήματα. Η εξάλληψη της φτώχειας ε, δεν πρόκειται να γίνει μέσα από ένα μαγικό μέτρο και να μην ξεχνάμε και τις επιπτώσεις της ε, τρέχουσας κρίσης. Ας ε, ενώσουμε τα χέρια για να επιτύχουμε ένα μίνιμουμ διεθνής συμφωνίας. Ο Σνάλφος Λούκας, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος στην Εστονία. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ενδέχεται να πρέπει να συστήσουμε νέους θεσμούς, οι ρυθμιστικές αρχές. Το θέμα είναι ότι στην Ευρώπη οποτεδήποτε ε, συστήνεται κάτι καινούριο, προκύπτει και η συνακόλουθη ε, γραφειοκρατία και τίνουμε να έχουμε περισσότερους υπαλλήλους από ουσία. Όσον αφορά στη διεθνή συνεργασία, Ένα δικαστήριο, ένα περιβαλλοντικό δικαστήριο ε, θα ήταν ίσως το σημαντικότερο. Όχι μόνο για να εγγυάται την εφαρμογή των κανονισμών που έχουμε θεσπίσει, αλλά και για να περιοριστεί η υποκρισία σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως όταν μιλάμε για την αντιμετώπιση της ε, υπερθέρμανσης του πλανήτη ή για τη μετάβασή μας ε, προς την πράσινη οικονομία πρέπει να αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση. Από την άλλη οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε τακτοποιήσει τα του οίκου μας. Όταν δηλαδή παράγουμε ενέργεια στην Ευρώπη, να σεβόμαστε το περιβάλλον. Οποτεδήποτε όμως εισάγουμε ενέργεια, παραδείγματος χάρη από τη Ρωσία, ε, τότε δεν διστάζουμε να εισάγουμε ενέργεια η οποία παρήχθη από την καταστροφή του περιβάλλοντος. Άλλο παράδειγμα, η εξαγωγή αποβλήτων από την Ευρώπη σε χώρες του τρίτου κόσμου συλλέγονται εδώ τα απόβλητα και εξάγονται σε χώρες του τρίτου κόσμου. Ε, αυτό είναι υποκρισία και δεν πρέπει να υπάρχει. Και τέλος, η κρίση είναι κάτι το ε, δυσάριστο, αλλά το να ξετύχει κανείς από την κρίση είναι πολύ πιο δύσκολο οι παραγωγοί, οι κατασκευαστές ε, αυτοκινήτων περιμένουν να κατασκευαστούν νέα μοντέλα και υπάρχει μια τεράστια αναμονή στην κατασκευή αυτοκινήτων ε, για το μέλλον. Ο Άλφος Ρόλι, πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Η κυρία Ρόλι. Ευχαριστώ. Σημαντική αυτή η συνάντησή μας. Από πλευρά Νομένου Βασιλείου, τα εξή. όλα τα εθνικά κοινοβούλια να μπορούν να αξιοποιήσουν τη χρονική περίοδο από τώρα μέχρι τον Ιούνιο για να αυξήσουν τη συνειδητότητα, την ενημέρωση του κοινού για το Ρίο και των ηγετών, ούτως ώστε οι ηγέτες μας να βοηθήσουν την συμβολή της Ένωσης για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο Ρίο. Μας ανησυχεί πολύ ότι ο δικός μας Πρωθυπουργό δεν έχει ακόμη δεσμευτεί ότι θα μεταβεί στο Ρίο το δεύτερο. Καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει την ισχυρότερη δυνατή διαπραγματευτική θέση και να δούμε πώς μπορούμε να συζητήσουμε με την κολομβιανή αντιπροσωπεία το θέμα των, της αηφόρων ανάπτυξης και των αηφόρων στόχων, των στόχων βιωσιμότητας μέχρι τον Ιούνιο. Και να τονίσω τη σημασία του ρόλου των κοινοβουλευτικών. Συμφωνώ με την ε, Γαλλίδα συνάδελφο. Πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της εκπαίδευσης και της αύξησης της συνειδητότητας των περιβαλλοντικών θεμάτων δεν είναι κατανοητά στο βαθμό που θα έπρεπε. Ενώ οι Υπουργοί Οικονομικών μας που ασχολούνται με την οικονομία χωρίς να λαμβάνουν υπόψη θέματα αηφόρου ανάπτυξης. Σας καλώ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι από τα διάφορα κοινοβούλια να δείτε πώς ε, μπορείτε στις χώρες σας να αυξήσετε τη συνειδητότητα. Πρέπει να υπάρξει πίεση από την κοινή γνώμη, από τα έξω, που να πιέζει όχι μόνο τους, βουλευ... τους υπουργούς, αλλά και τους ίδιους τους βουλευτές, ούτω ώστε να δεσμευθούν να υπάρξει η δυνατότερη, ισχυρότερη δυνατή διαπραγματευτική θέση. Πρέπει να δούμε και τα θέματα που αφορούν όχι μόνο τη δική μας γενιά, αλλά και τις επόμενες. Είναι πολύ σημαντικό και σας καλώ όλους να εργαστείτε και να δεσμευτείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ ο συνάδελφο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συνάδελφο, η κυρία Κούκοβιτ. Σα ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ρίο αποτελεί την ε, ευκαιρία να δώσουμε μία απάντηση στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση. Μπορούμε ε, προβάλλοντας την βιώσιμη ανάπτυξη και αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της ε, λειψιδρίας. Αυτά μοιάζουν με ασθενή, με χρόνια ασθένεια. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να κινούμαστε διαφορετικά, να διατρεφόμαστε διαφορετικά. Ε, όπως ακριβώς συμβαίνει και όταν, όπως σας είπα, καλείται κανείς να αντιμετωπίσει μία ασθένεια. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση και με τον τρόπο αυτό οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και την ε, έλλειψη πόρων. Ε, χρειαζόμαστε ανάπτυξη για να απασχολήσουμε τους νέους όμως ε, πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση των πόρων. Ανάπτυξη με περιορισμό πόρων, αυτό είναι δύσκολο και ίσως και να μην είναι και λογικό. Πρέπει όμως να το πράξουμε αυτό και πρέπει να το επιβάλλουμε και μέσα από τη σχετική νομοθεσία και με την ευαισθητοποίηση των πολιτών ε, στην βιώσιμη ανάπτυξη, μεγάλη ευκαιρία θα έχουν οι καινοτόμε επιχειρήσεις, τα ρηξικέλευτα προγράμματα. Αυτά συμπεριλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα Horizon 2020. Ε, ε, για να γίνουν όλα αυτά, ε, χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Χαιρετίζω τη σημερινή συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την κρίση και να προβάλλουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστούμε κυρία Κουκουμπίτς για αυτή την ε, εύληπτη εικόνα, την ανάγλυφη εικόνα και την, την παρομοίωση με τον ασθενή. Τώρα λοιπόν έχουμε ε, τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, του Λουξεμβούργου, συνάδελφος κ. Μπόντεμ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ε, οργάνωσε αυτήν την ενδιαφέρουσα ε, συνεδρίαση και οι προλαλήσαντες ε, επέμειναν στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην διάσκεψη Ρίο συν 20. Ζήσαμε στην Κοπενχάνη, ε, Κοπενχάγη μια ε, κακοφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μηνύματα που προέκυψαν κάπως αντίξωα στο Τυρμπάν ε, υπήρχε ε, ως βασικός διαπραγματευτής ε, πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι καταφέραμε να πιέσουμε, να υποχρεώσουμε όσους δεν ήθελαν να προχωρήσουν να κάνουν περισσότερα από όσα ήθελαν πριν από την διάσκεψη. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να παίξουμε έναν ρόλο καταλήτη στο Ρίο συνήκωση Υπάρχει ο κίνδυνος ε, στο ε, Ρίο να ε, υπάρχουν πολύ, να παρίστανται πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια κακοφωνία μηνυμάτων. Γι' αυτό κατά τη γνώμη μου το καλύτερο θα ήταν να επικεντρωθούμε στο ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, ο οποίος πρέπει να αποστείλει ένα μήνυμα με μεγαλύτερη συνοχή. Κάποιες ε, ανάπτυξη χώρες θέλουν να κάνουν περισσότερα από ό,τι άλλες, πρέπει όμως ε, εμείς να τηρήσουμε τις υποσχέσεις ε, που τους δώσαμε πριν από 20 χρόνια. Υποσχεθήκαμε πολλά πράγματα, όμως δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις αυτές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το εξής. Η αναπτυξιακή βοήθεια, για παράδειγμα. Είπαμε 7% του ΑΕΠ ε, να πάει στην αναπτυξιακή βοήθεια. Πόσες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κάνουν αυτό. Νομίζω 0,7% συγγνώμη, νομίζω ότι είναι ε, πολύ σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο για την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Ελπίζουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες δράσεις, ε, σε μετρήσιμους ε, ε, στόχους και είναι σημαντικό επίσης να ενισχύσουμε το πρόγραμμα του ΟΗΕ για το περιβάλλον. Πολλοί το είπαν αυτό, κατά τη γνώμη μου. Το είπε και ο Γιώ να, πρέπει να έχουμε ένα συμβούλιο ε, αηφόρου ανάπτυξης που παρακολουθεί ότι οι υποσχέσεις ε, που ε, δίνονται και οι στόχοι που τίθενται πράγματι εκπληρώνονται. καλό θα ήταν να καταλήξουμε και σε έναν δίκτυ ευημερία ε, που θα συμπληρώνει το ε, ΑΕΠ. Και αν έχουμε έναν τέτοιο δίκτυ σε διεθνές επίπεδο αναγνωρισμένο, νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο οι στόχοι της αηφόρου ανάπτυξης ε, και να επιτευχθούν και να είναι πιο μετρήσιμοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος από τη Τβέιντε Κάμερα, ο συνάδελφος Φαντιβέρτ. Ή συνάδελφος Φαντιβέρτ. Ευχαριστώ για τη συνάντηση αυτή σήμερα. Σήμερα στην ε, Ολλανδία έχουμε τη γιορτή του δέντρου με την οποία προσπαθούμε να έχουμε μια μικρή συμβολή στην βιοπικιλότητα. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε λοιπόν στο Ρίο οικονομία και οικολογία, τι πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε και τους δύο τομείς. Για να υπάρξει μια κοινή στάση για την ε, πράσινη οικονομία χρειάζεται να παίξει το ρόλο του και ο κόσμος της οικονομίας και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η Ολλανδία θέλει να υπάρξουν συναντήσει μεταξύ τη πολιτική και τη οικονομία για τον τομέα αυτό. Επίση, μιλήσαμε για ένα χάρτη πορεία. Βεβαίω, υποστηρίζουμε αυτή την ιδέα, θα μα επιτρέψει να καθορίσουμε και στόχου και τα μέσα. Και όταν μιλάμε για μέσα δεν είναι μόνο νομικά και οικονομικά μέσα και εργαλεία. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία τη οικονομική και κοινωνική πολιτική Προγράμματα μαθητεία, για παράδειγμα είναι πολύ σημαντικά για την πράσινη οικονομία. Και τρίτον, η πράσινη διακυβέρνηση και αυτή σημαντική. Συμφωνώ με τις εκκλήσεις που έγιναν για να ενισχυθεί το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον. Υπάρχει κρίση σε πολλούς τομείς, άρα χρειάζεται σφαιρική αντιμετώπιση επίσης. Αυτό θα είναι ουσιαστική πρόοδος. Και κυρίως να σκεφτόμαστε ε, τοπικά αλλά και να δρούμε τοπικά. Ευχαριστώ. Ο κ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας ε, να συναντιόμαστε σήμερα με τους ε, συνάδελφούς μας, τους βουλευτές ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων για τα ζητήματα Ρίος συνένα εδώ και 20 χρόνια, μετά από το Ρίο ε, του 1992, μετά το Johannesburg ε, ε, και μέχρι το, τον Ιούνιο, να δούμε ποιες πρόοδους, τι πρόοδο έχουμε, έχουμε σημειώσει και να δούμε επίσης ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που πρέπει να έχουμε εν ώψη του, της διάσκεψης τον Ιούνιο. Πρώτο σημείο που θα ήθελα να θίξω, ε, το είπε ο συνάδελφος Κερβάντη, υπάρχει ένα πρόβλημα διακυβέρνησης σε επίπεδο ΙΕ. Πρέπει λοιπόν η σύνοδη κορυφή μας να μην ε, είναι απλώς σπαρμένες με καλές προθέσεις, αλλά να ε, υπάρχει ένας ρεαλισμός, τα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της κοινή γνώμης και τη καθημερινή ζωή τη. και γι' αυτό νομίζω ότι το κείμενό μας ε, είναι ε, ένας ενδιαφέρον τρόπος να το πετύχουμε. Κάτι ακόμη... Επειδή ε, ήμουν πριν από τρία χρόνια στην Κοπενχάγη μαζί με άλλους συναδέλφους, δεν είναι δυνατόν ε, να υπάρχει αυτή η ε, διαφορά ανάμεσα στην κοινή γνώμη και ε, στους κυβερνώντες. Τρίτον, πρέπει να υπάρχει μια αξιοπιστία σε σχέση με τα ζητήματα της αηφόρου ανάπτυξης και νομίζω ότι είναι ένας αγώνας που πρέπει να δίνουμε συνεχώς ε, με την ευκαιρία μιας τέτοιας διάσκεψης ε, για το θέμα της κλιματικής αλλαγής για παράδειγμα 250.000 πρόσφυγες κλιματικοί ε, υπάρχουν και είναι ένας αριθμός που θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο μέχρι το 2050. Αυτό το πράσινο αυτό το πράσινο ταμείο ε, το οποίο αποφασίσαμε στο, ε, στο Ντριμπάν ε, να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί 100 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν στις βιομηχανοποιημένες χώρες μέχρι το 2020 για να εξαλειφθεί η φτώχεια και να υπάρξει μια πολιτική ανάπτυξη. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που θα συζητηθούν και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ο συνάδελφος Όλακ από το Πολωνικό Κοινοβούλιο. Η συνάδελφος είναι αντιπρόεδρος της ε, ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε τους ε, οικολογικούς στόχους αλλά και τους ε, κοινωνικούς και αυτό είναι η χάραξη μιας ε, πολιτικής η οποία προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και σε τομείς που έχουν σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, καταρχήν ε, πρέπει να δούμε λιγάκι τα επιτεύγματά μας ε, στον τομέα αυτό, να κάνουμε έναν έλεγχο. Αυτό πρέπει να γίνει από αρμόδιους φορείς και πανεπιστήμια. Εξάλλου είναι σημαντικό να επηρεάσουμε λιγάκι τις επιθυμίες των πολιτών, δείχνοντάς τους δηλαδή ότι και οι ίδιοι μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον, κυρίως ε, με τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν για τις καθημερινές τους αγορές. Βεβαίως, ε, εξίσου σημαντική είναι και η προαγωγή της ε, κοινωνίας των πολιτών, η δημιουργία μιας περιραίουσας ατμόσφαιρας ε, που θα ευνοεί ε, τη σωστή τοποθέτηση απέναντι στη βιωσιμότητα. Και εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριος Μέρκες και μετά ακολουθεί ο κύριος, ε, η κυρία και μετά ακολουθεί ο κύριος Πρόντι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για αυτή τη μοναδική συνάντηση που γίνεται σήμερα στο Κοινοβουλίο και το Ρίο θα είναι μια μοναδική ευκαιρία. Ε, απευθύνομαι κυρίως ε, στους συναδέλφους από την Δανία Think Global and Act Global. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το Ρίο αφορά το μικροεπίπεδο διότι ήδη έχουμε τόσα πολλά παγκόσμια γεγονότα που αφορούν την μακροοικονομία, τη μακροπολιτική. Εδώ όμως μιλάμε για θέματα που αφορούν ε, την καρδιά των ανθρώπων. Ε, πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε όλους ε, για το πού κατευθύνεται η γη. Το άλλο θέμα που θέλω να δείξω γιατί συμφώνησε ότι θα είναι παρόν και ο κύριος Μπαρόζο. Ρωτώ, θα είναι παρόν ο Δανός πρωθυπουργός. γιατί νομίζω ότι αυτό θα ε, βελτιώσει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν είναι σημαντικό να είμαστε συγκεκριμένοι, να συζητήσουμε για το νομοθετικό πλαίσιο. Όσον αφορά τους, τις πρώτες ύλες βλέπουμε ότι κατευθυνόμεθα προς ε, μια ε, βελτίωση τόσο στις Ηνωμένε Πολιτείε όσο και σε σχέση με την επικείμενη οδηγία περί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βεβαίως ε, αυτά αφορούν και πάλι τα σκληρά οικονομικά, τη ροή των πρώτων υλών. Δεν πρέπει όμως, ε, πρέπει να ασχοληθούμε και με τη διαφάνεια, με το τι ακριβώς γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Τι παράγεται, ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό λοιπόν θα πρέπει, είναι ένα από τα θέματα στο Ρίο, έτσι ώστε να συζητήσουμε μια πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Γιατί πρέπει να καταλήξουμε σε μια οικονομία με μηδενικά απορρίμματα ε, και νομίζω ότι η διαφάνεια θα βοηθήσει. Να πω λοιπόν ότι ε, τη χρονιά του blueprint για το νερό που θα έρθει σύντομα είναι σημαντικό να συζητήσουμε το νερό. Γιατί ένα πράγμα είναι σαφές ε, ότι στην οικονομία μας, όπως είναι προγραμματισμένη για το μέλλον, δεν θα υπάρχει ε, ο αγώνας ανάμεσα στη γη ε, και ε, τα, τις πρώτες ύλες που βασίζονται σε βιολογικές ενέργειες. Το βασικότερο που θα προκύψει στο μέλλον θα είναι το πρόβλημα του νερού. Επόμενος είναι ο κύριος Πρόντι και μετά ο κύριος Επιρέλου. Βιτόριο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινώ πρώτα απ' όλα από τη διαπίστωση ότι είναι ε, πεπερασμένη η φυσική πόρη ε, βλέπω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο για τους ε, φυσικούς πόρους ε, να υπάρχει το δικαίωμα του ανθρώπου, το οποίο προστίθεται στον κατάλογο των ανθρωπίων δικαιωμάτων, το δικαίωμα του ανθρώπου στην πρόσβαση στους φυσικούς πόρους. Γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αλεξάρτησης. Ήδη τώρα Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση της αλληλεξάρτησης. Κατόπιν τούτου οφείλουμε να βρούμε τον τρόπο να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά αυτή την αλληλεξάρτηση. Και βλέπω λοιπόν ότι εδώ είναι απόλυτα απαραίτητο να ε, μεταρρυθμιστούν οι διεθνείς ε, θεσμοί, ε, ξεκινώντας βέβαια από τα Ηνωμένα Έθνη, που τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνες και για οργανισμούς του Bretton Woods, αλλά και για άλλους οργανισμούς, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Αυτά σας τα λέω για να μην ξεχνάμε, όπως σας είπα, ότι έχουμε πεπερασμένους πόρους. Αλλά χρειάζονται και συγκεκριμένες δράσεις, έτσι ώστε η κοινωνία μας να απελευθερωθεί από τον ηλισμό. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κατανοήσουμε είναι πώς μπορούμε και πρέπει να επενδύουμε σε άτομα και στις ικανότητες των ανθρώπων να συμπεριλαμβάνονται στη διαχείριση των θεσμών, σε όλα τα επίπεδα. Το τελευταίο που θέλω να υπογραμμίσω είναι το εξής. Να, ε, σας, να πω πόσο επιγόντως απαραίτητο είναι να υπάρξει και κάτι άλλο. Η έννοια του δημόσιου αγαθού, του κοινού αγαθού μάλλον. Αυτό το έχουμε ήδη αναφέρει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε έναν άλλο τρόπο να ξεφύγουμε ως κοινωνία από τα υλικά αγαθά. Ευχαριστούμε. Επόμενος ο κύριος Πιρέλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που όλοι μοιάζουμε να έχουμε την ίδια γνώμη όσον αφορά τους στόχους που θέλουμε να υπερασπιστούμε, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Να εκφράσω την ανησυχία μου, γιατί στο πλαίσιο στο οποίο θα γίνει αυτή η συνάντηση κορυφής, το πλαίσιο αυτό είναι η διεθνής, η παγκόσμια οικονομική κρίση που προκαλεί τεράστιες περιχοπές. Άλλες δικαιολογημένες και άλλες όχι. Αυτό ε, δεν θα βοηθήσει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και δεν θα βοηθήσει την αηφόρο ανάπτυξη. Παράδειγμα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μειώσει τις εκπομπές, για παράδειγμα, στο εναέριο χώρο, κάποιες άλλες χώρες μας ε, απειλούν με πολύ σκληρές οικονομικές ε, κυρώσεις. Αυτό δεν πρέπει να το δεχτούμε. Εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες, αλλά οι κυβερνήσεις υφίστανται πιέσεις από τις πολυεθνικές και τους κλάδους βιομηχανίας. Πιστεύω ότι ο πειρασμός να μην συνδυάσουμε την οικονομική με την οικολογική διάσταση λόγω της κρίσης είναι υπαρκτός. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν τα κοινωνικά μέτρα να μην εφαρμόζονται, κοινωνικά μέτρα που επίσης έχουν οικολογική διάσταση. Χωρίς την κοινωνική διάσταση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη, ό,τι και να πούμε ότι υπερασπιζόμαστε το περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν ως βουλευτές πρέπει να επαγρυπνούμε ιδιαίτερα διότι εάν οι προηγούμενες ε, συναντήσεις κορυφής δεν ήταν ικανοποιητικές, τώρα που έχουμε την κρίση που αξιοποιείται ως πρόσχημα για πολλά άδικα μέτρα, εδώ λοιπόν θα έχουμε ακόμη περισσότερες δυσχέρειες. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε αυτούς που λένε ότι πρώτα θα αντιμετωπίσουμε την κρίση και μετά το οικολογικό πρόβλημα. Όχι, οι προτάσεις μας πρέπει να στοχεύουν στο συνδυασμό της αντιμετώπισης οικονομίας και οικολογίας. Ευχαριστώ. Ο Σνάλφος, Πίσοφο Πύλος και μετά Ρόσμπαχ και Χίπνα. Και ε, θα έχουμε λοιπόν δώσει το λόγο σε όλους όσους τον ζήτησαν. Παρακαλώ. Ο Σνάλφος, Χρυσόγελος, Σνάλφος Χρυσόγελος. Δεν είναι παρόν ο συνάδελφος Χρυσόγελος. Άννα Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ε, καλωσορίζω όλους όσους είναι εδώ και να ευχαριστήσω τον επικεφαλής της, ε, τον εκπρόσωπο της Δανέζικης ε, Προεδρίας. Ήμουν και εγώ στην Κομεχάγη και το πρόβλημα νομίζω είναι ότι τα εθνικά συμφέροντα είναι τόσο διαφορετικά, αλλά και οι ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν οι συναντήσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές, όπως αυτή που κάνουμε εδώ, για να καταλάβουμε τις ανάγκες ημέν των δε. Οι περισσότερες χώρες του τρίτου κόσμου θέλουν φυσικά οικονομική στήριξη. Δυστυχώς όμως δεν είναι εύκολο να χορηγηθεί. Εάν θέλουμε να αξιοποιήσουμε ε, τις πιστώσεις και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τεράστια ποσά στη διάθεσή μας, πρέπει τα χρήματα αυτά να δαπανηθούν για πολύ συγκεκριμένα προγράμματα και να ξέρουμε τι αποτελέσματα θα έχουμε. Στην Ευρώπη έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για να αξιοποιήσουμε τους πόρους μας. Ένα μικρό παράδειγμα. πηγαίνουν τα σκάφη μας και αλλιεύουν στις χώρες τρίτου κόσμου, στα ύδατα των χωρών τρίτου κόσμου. Ενώ από την άλλη πλευρά στις χώρες μας ε, πολλά τρόφιμα καταλήγουν στα σκουπίδια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους δικούς μας πόρους και να βοηθήσουμε έτσι και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Να τα βγάλουν πέρα μόνες τους με βάση τις δικές τους πηγές. Να γίνουν περισσότερο αυτάρκεις. Επίσης, ορισμένοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο θέμα της καταστροφής των δασών που έχει τεράστιες επιπτώσεις στο κλίμα μας διότι είναι εξέφρενη η αποψήλωση των δασών. Στην Ευρώπη έχουμε τις αναγκαίες υποδομές για αναδάσωση. Θα έπρεπε αυτή μας την πείρα να την περάσουμε και στις τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε στον κύριο Χρυσόγλου που τον είδα προηγουμένω. Ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ένα ηγετικό ρόλο στην ε, διάσκεψη για το Rio 20, αλλά πρέπει να το κάνει αυτό με δύο τρόπους. Μέσα από, δεσμευτικές, μέσα από δεσμεύσεις και στόχους που θα προωθήσει, αλλά ταυτόχρονα και μέσα από μια στρατηγική που θα οδηγήσει σε πλειοψηφία στη συνδιάσκεψη, έτσι ώστε να υποστηριχθούν ενεργά αυτοί οι στόχοι έχοντα την εμπειρία από τη συνδιάσκεψη στα 10 χρόνια που έγινε στο, στο Johannesburg το, το 2002, πιστεύω δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη από την αδύναμη παρουσία τότε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την απουσία μια κοινή στρατηγική και δεσμευτικών στόχων, που μπορούσε να έχει οδηγήσει σε απογοητευτικά αποτελέσματα αν δεν υπήρχε την τελευταία στιγμή η μεγάλη πίεση τη κοινωνία των πολιτών για να διασώσει τα αποτελέσματα. Κατά βάση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ένα ισχυρό ηγετικό ρόλο και πριν τη συνδιάσκεψη, όχι μόνο περιμένοντας στη διάρκεια της συνδιάσκεψης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία του και με άλλα εθνικά κοινοβούλια, να μην περιοριστεί μόνο στα κοινοβούλια των κρατών μελών, αλλά αξιοποιώντα τι συνεργασίε του και τι σχέσει του με άλλα κοινοβούλια εκτό Ευρώπη, να μπορέσει να επηρεάσει τη διαδικασία πριν. Και επίση νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ σημαντική και ισχυρή η παρουσία τη κοινωνία των πολιτών και τη αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε πραγματικά η κρίση που υπάρχει σήμερα να μην είναι η αφορμή για να ε, απεμπολιστούν οι στόχοι της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής, αλλά αντίθετα να ενδυναμώσει και να, υπάρξουν, να ενδυναμώσει η κίνηση και να υπάρξουν δεσμεύσει για κοινωνική συνοχή, αντιμετώπιση φτώχεια, προστασία του κλίματο, στροφή στην πράσινη οικονομία και δημιουργία θέσεων απασχόληση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Η συνάδελφο Χίμπνα. Εδώ και 20 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε ανακεφαλαίωση των ε, αποτελεσμάτων, ε, τι επιτύχαμε στο παρελθόν και τι προσδοκούμε για το μέλλον. Όμως, για να προβούμε σε απολογισμό, καταρχήν θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα τι ακριβώς εννοούμε με την έννοια βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλιώς το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι στην Αφρική και αλλιώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διευκρινιστεί ε, ποιοι είναι οι παράγοντες ε, που συμπεριλαμβάνονται στη βιώσιμη ανάπτυξη ε, και κυρίως όσον αφορά βιώσιμη ανάπτυξη Αφρική και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι και τα κριτήρια που συγκρίνουμε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι κάτι που μπορεί κανείς να το βλέπει, να το εξετάζει στο σύνολό του ή μπορεί να το αντιμετωπίζει ως ε, το άθροισμα πολλών ε, παραγόντων ε, στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης σε διάφορες χώρες. Με την καινοτομία με ε, σύγχρονες υπηρεσίες καινοτόμα προϊόντα, νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο. Όλα αυτά όμως δεν είναι εφικτά χωρίς ε, να προάγεται παράλληλα και ο κοινωνικός διάλογος. Μόνο με τη συμπερίληψη της κοινωνίας θα καταστεί δυνατόν να βρούμε λύση. Χωρίς το διάλογο, χωρίς την ολοκλήρωση στο κατώτατο επίπεδο, χωρίς την κοινωνική αποδοχή, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Και ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η ενέργεια. Η αντιμετώπιση της πυρηνικής ενέργειας, η μη αποδοχή της από πλευράς πολιτών. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να καταλήξουμε σε ισορροπία. Πρόεδρος. Όλο... Ευχαριστώ. Έτσι κλείσαμε το κατάλογο μιλητών. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Λόκλιν που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δανέζικου Κοινοβουλίου για να κάνει μια καταληκτική ομιλία και κατόπιν ε, ε, είστε όλοι καλεσμένοι σε ένα μεσημεριανό γεύμα συζήτηση όπου σας καλεί ο πρόεδρος Μάρτιν Σούλτς του Κοινοβουλίου όπου θα έχουμε δυνατότητα να συνεχίσουμε να συζητάμε. Είστε όλοι ιδιαίτερως ευπρόσδεκτοι στις μία ώρα. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύ ενεργό συμμετοχή σα στη συζήτηση. Νομίζω η συζήτηση που είχαμε ήταν πάρα πολύ καλή και επίση από τη συζήτηση κατέστη σαφέ ότι όλοι θυμόμαστε πάρα πολύ καλά το Ρίο του 92. Τον ενθουσιασμό που νιώθαμε τότε για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε, να δεχτούμε ότι μέχρι τώρα δεν επιτύχαμε πολλούς από τους στόχους που είχαμε θέσει τότε. Η συζήτηση για το πώς ε, μπορούν να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Επ' αυτού η κυρία Γόλης από το Ηνωμένο Βασίλειο πολύ σωστά επισήμανε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, θα συνειδητοποιήσουν οι δικοί μας οι πολίτες το τι ακριβώς συμβαίνει ε, και να ε, προσπαθήσουμε να τους εμφυσίσουμε ενθουσιασμό. Η παιδεία είναι πολύ σημαντική, όπως ήταν και στις αρχές της δεκαετίας των 90, τότε όταν είχαμε την Agenda 21 που και αυτή θελήσαμε να την προάγει η κοινωνία των πολιτών. Βεβαίως και πρέπει να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους μας, τους βουλευτές και με τις κυβερνήσεις. Εγώ εκπροσωπώ ένα από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού στην πατρίδα μου και εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα για τα θέματα, συμφωνούμε όλοι από αυτόν. Αλλά και πάλι όσον αφορά τη συνδυάσκεψη στο Ρίο είναι σημαντικό να έρθει ο ε, Πρωθυπουργός ε, ή Πρωθυπουργό της ε, Δανίας ε, να παραβρεθεί στο Ρίο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό η Πρωθυπουργό να προάγει την ατζέντα αυτή σε ολόκληρο τον κόσμο. κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μεγάλα βήματα, όχι μικρά. Εδώ και 20 χρόνια κάνουμε μικρά βήματα. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να κάνουμε μια ριζική αλλαγή, η αλλαγή αυτή να έρθει από κάτω προς τα πάνω, οι κυβερνητικές δομές να είναι πιο αυστηρές και με μεγάλο ενδιαφέρον ακούσαμε αυτά που είπατε για το αντεχόμενο του ποινικού δικαστηρίου. Ένα σύστημα παρεμφερές με αυτό του ΠΟΕ που όπως είπατε ε, θα μας βοηθήσει να μην είμαστε υποκριτές ε, όταν αγοράζουμε κυρίως ενέργεια από το εξωτερικό. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, να συμπεριλάβουμε και την επιχειρηματική κοινωνία την ατζέντα ε, ε, CSR να τη συμπεριλάβουμε στις διαπραγματεύσεις μας. Επίσης, ε, η ατζέντα μας για το CSR να είναι δεσμευτική, έτσι ώστε να επιτύχουμε πρόοδο. Λυπάμαι που δεν μπορώ ε, να ε, συμπεριλάβω την ε, εισήγησή μου όλα αυτά που ελέγχθησαν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη είμαστε σε προνομίου θέση. Έχουμε το καθήκον να αλλάξουμε το σύστημά μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συνδιάσκεψη του Ρίο έχει σχέση ε, και με τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στον κόσμο, ε, με τη φτώχεια που βλέπουμε σε πολλές χώρες, όχι μόνο στις λιγότερο αναπτυγμένες. Είναι λοιπόν σημαντικό να προβάλλουμε και το στόχο του 0,7% βοήθεια ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες η δική μου χώρα συμμετέχει σε αυτό, αλλά και όλες οι υπόλοιπες χώρες πρέπει να βοηθήσουν να υπάρχει καλύτερος καταμερισμός, έτσι ώστε η βιώσιμη ανάπτυξη να ε, υπάρξει παντού. Επ' αυτού χρειαζόμαστε συγκεκριμένους στόχους και νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε και τους στόχους της χιλιετίας που νομίζω προέβαλε η Κολομβία. Φαντάζομαι ότι όταν θα επιστρέψετε στις πατρίδες σας θα συνεχίσετε αυτή τη συζήτηση και θα ασκήσετε πίεση στους ηγέτες της χώρας σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και που μου δώσετε με την ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο. Πρόεδρος, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον μείγμα. Ε, ένα μείγμα το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε παντού, στις κυβερνήσεις, σε όλες ε, τις ευκαιρίες. Αυτό που μας ισχύει περισσότερο είναι σχετικά με το Ρίο δεν είναι σαφής ε, η θέση μας. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε μια πολύ καλή αρχή έτσι ώστε να ξεκινήσει η επικοινωνία στα 27 κράτη-μέλη. Ε, αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ήρθατε εδώ σήμερα. Σας εύχομαι καλή όρεξη και ε, θα ξεκινήσουμε και πάλι στις 3 με το δεύτερο τμήμα των συζητήσεών μας θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ποτόσνικ ως κύριο Μιλτή, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και μετά θα έχουμε και πάλι τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Καλή σας όρεξη. Γεια σας.